Uh, Συνάδελφοι, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε, η κυρία Βαλεάν αποσιάζει, οπότε πρέπει εγώ να την αντικαταστήσω. Και έχουμε δύο προσκεκλημένους ε, σήμερα. Στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης καλωσορίζω τον κύριο Αλμπέρτο Ποντότσνικ και την Κλάρα Πολέτη που είναι υπεύθυνη του του κανονισμού ΆΣΕΡ και του ε, αρμόδιου οργανισμού. Ε, μιλάμε για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και για αυτό το στόχο ο οργανισμός προετοιμάζει μια ετήσια έκθεση εποπτείας της αγοράς και μιλάμε για όγκους ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ε, σε, ε, στην χονδρική πώληση. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ΆΣΕΡ ε, πρέπει να υποβάλλεται το σχέδιο προγράμματος εργασίας ετησίως. Έχουμε λοιπόν μία ώρα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ποτόζη και στην κυρία Πολέτη για να μας παρουσιάσουν την ετήσια αυτή έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Πάντοτε ε, με χαρά επισκέπτομαι την Επιτροπή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι όμως η τελευταία γιατί η θητεία μου λύγει στα τέλη του έτους και μετά θα έρχεται εδώ ο διαδοχός μου. Είμαι λοιπόν ε, ε, πολύ ικανοποιημένος που είμαι σήμερα εδώ για να σας παρακολουθήσω την έκθεση εποπτείας της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο ώστε να αφήσω όσο γίνεται ε, περισσότερο χρόνο σε εσά για να συζητήσουμε ε, το θέμα. Πρόγραμμα εργασίας λοιπόν, αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε ένα σχέδιο προγράμματος εργασίας, καταρχάς γιατί αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί όταν θα υιοθετηθεί ο προπολογισμό της Ένωσης. Ετησίως υποβάλλουμε πρόγραμμα το οποίο είναι σύμμορφο προς το αίτημά μας για πόρους και είμαι πάντοτε ευγνώμων στην Επιτροπή Ίδρυ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πάντοτε στηρίζουν τα αιτήματά μας για επιπλέον πόρους και προσωπικό. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, γνωρίζετε ποια είναι η υπόθεση, ποια είναι, πώς πάει. Ε, κάποιες φορές παίρνουμε παραπάνω πόρους, κάποιες όχι. Πιθανότατα, ελπίζω πως αυτό δεν θα αλλάξει, αλλά ε, πιθανότατα περιμένουμε και την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και ε, στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις. Τώρα, εμείς συντάσσουμε το, πρόγραμμα, το σχέδιο προγράμματος εργασίας με αναφερόμενοι σε έξι ειδών δραστηριότητες. Έχουμε το πολιτική με, ε, για, με βάση τον κανονισμό για την εσωτερική αγορά και τη διαφάνεια, που εστιάζουμε στα συστήματα που στηρίζουν την εργασία του οργανισμού για την ακερότητα της αγοράς και τη διαφάνεια. Δεύτερος πυλώνας είναι η εποπτεία της αγοράς και η ιδεοντολογία. Εκεί προσπαθούμε να καταγράψουμε τα αποτελέσματα της εποπτείας μας. Δηλαδή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε οποιοδήποτε περιστατικό ακατάλληλη συμπεριφορά στην αγορά και έπειτα να κοινοποιήσουμε στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή ε, στις αρχές ε, επιβολής του νόμου για ύποπτες ε, καταστάσεις στην αγορά. Μετά έχουμε τη δραστηριότητα υποπτές της αγοράς που σας παρουσιάζω σήμερα τα αποτελέσματα. Ε, θα σας τα δώσω με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Έχουμε την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου που αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε το τρίτο πακέτο καθαρής ενέργειας και των, δικτύ... και των ε, κωδικών του δικτύου, γιατί ξέρετε ότι στην ηλεκτρισμό έχουμε διάφορους όρους, προϋποθέσεις και μεθοδολογίες και είμαστε στο στάδιο υιοθέτηση αυτών. Αυτά είναι τα κλειδιά για την ε, ε, ορθή λειτουργία του συστήματος. Και τέλος, δουλεύουμε και στον τομέα των υποδομών και της ασφάλειας των εφοδιασμού πράγμα που έχει να κάνει με την συμμετοχή μας στην ανάπτυξη του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης δικτύων του ορισμού των project κοινού, κοινής ωφελίας και επίσης ε, πώς τα διασυνοριακά προγράμματα ε, είναι όντως διασυνοριακά και εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις για την υλοποίησή τους. Δεύτερο, η διαφάνεια είναι ο κατάλογος με νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον οργανισμό μας μετά από το, πακέτο, το νέο πακέτο για την ενέργεια. Αυτά όλα θα εφαρμοστούν το πακέτο της καθαρής ενέργειας. Το γνωρίζετε γιατί είναι η νομοθεσία που εσείς περάσατε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ορισμένα από αυτά τα ζητήματα είναι πολύ επίμαχα και περίπλοκα. Και είναι πολύ σημαντικά για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την ανεφοδιασμό ενέργειας για την Ευρώπη. Είναι κάτι, λοιπόν, που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι, και επιπλέον ομπειρογνώμονες. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να συμφωνήσουμε ανάμεσα στους συνομοθέτες για αυτό το νομοθέτημα. Και τώρα το έργο αυτό έχει περάσει στον οργανισμό για να ορίσει τις λεπτομέρειες. Και όπως γνωρίζετε από τις μεθοδολογίες, οι λεπτομέρειες είναι οι δύσκολες. Και ελπίζω πως αυτό θα λειτουργήσει ε, ενισχύοντας την ανάγκη για επιπλέον πόρους, σύμφωνα με το δικό μας αίτημα. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω στην έκθεση περί υποπτίας της αγοράς που παρουσιάζει τα βασικά αποτελέσματα και μετά Εάν σας ενδιαφέρει, ε, ε, θα επανέλθω στο πρόγραμμα εργασίας. Η έκθεση, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, περιλαμβάνει τέσσερις ε, τόμους. Εδώ σε δέκα λεπτά, που έχουν γίνει 7, μπορώ μόνο να εστιάσω σε κάποια κύρια μηνύματα. Δεν θα δούμε την χειραφέτηση του καταναλωτή. Θα εστιάσουμε περισσότερο στις ε, πωλήσει ε, χονδρικής, όπου εκεί είναι η ουσία. Πρόκειται για μια έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με τους Ευρωπαίους ε, ρυθμιστές για την ενέργεια. Εδώ τα πρώτα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να μας αφορούν. Δηλαδή ποιες είναι οι τιμές που εμείς πληρώνουμε. Είδαμε λοιπόν το 18 μια αντιστροφή της δραστηριότητα. Έχουμε περιορισμό του κόστους, μείωση του κόστους και αυτό αντικατοπτρίζεται στο σύνολο του λογαριασμού που πληρώνουμε. Ο ηλεκτρισμός μειώθηκε από το 41% το 2012 στο 35% το 2017 και μάλιστα το έχω πει αρκετέ φορέ ότι ακριβώ εκεί οι ανταγωνιζόμενοι προμηθευτέ ε, σε αυτό το κομμάτι ανταγωνίζονται. Το γεγονό ότι αντιστρέφεται τώρα αυτή η τάση, τουλάχιστον το 2018, είναι καλό σημάδι για τον ε, ανταγωνισμό των προμηθευτών. Επίσης από αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε, αν δείτε τις δύο γραμμές, η κάτω γραμμή η κίτρινη είναι αυτή που ορίζει την τιμή χονδρικής και η πάνω γραμμή, η πράσινη, είναι η λιανική τιμή. Βλέπουμε πως αυτές οι δύο γραμμές δεν συμπίπτουν, δεν αντιστοιχούν μάλλον η μία στην άλλη. Σημαίνει ότι ο, τελευταίο, ο τελικός καταναλωτής δεν μπορούσε να ωφεληθεί από την μείωση της τιμής χονδρικής που παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται πως θα αλλάξει τώρα. αλλά θα δούμε αν η βελτιωμένη αυτή αντιστοιχεία θα επαληθευτεί τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό ήθελα να εστιάσω όσον αφορά την ε, αγορά αλλιανικής και αν θέλετε μπορώ να επανέλθω αργότερα τώρα. Για την αγορά φυσικού αερίου βλέπουμε μια βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και θα σας δώσω κάποια γραφήματα που το δείχνουν αυτό. Αν και το μέλλον φαίνεται να είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Έχουμε λοιπόν κατηγοριοποιήσει τις ε, χώρες ανάλογα με το επίπεδο ρευστότητας και το βαθμό της εύρυθμης Λειτουργία λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου. Όσο πιο σκούρη είναι η χώρα, τόσο πιο εύρυθμα λειτουργεί η αγορά φυσικού αερίου. Κάποιες χώρες έχουν βελτιώσει την ε, απόδοση της αγοράς χοντρικής ε, της χοντρικής αγοράς για φυσικό αέριο, όπως η Ισπανία, η Αυστρία, αλλά βλέπουμε και άλλες αγορές που δεν καταφέρνουν να αναδυθούν και να λειτουργήσουν. Αν δούμε όμως την ρευστότητα της μελλοντική και της προηγμένης αγοράς, βασικά μόνο δύο αγορές έχουν σημαντική ρευστότητα, δηλαδή η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που όπως βλέπετε χρωματίζονται και με πιο σκούρο μπλε. Υπάρχουν λοιπόν διαφόρων ειδών προβλήματα. Όμως αναζητούμε τη σύγκληση και στο κόστος πηγής, ε, δηλαδή ε, μάλλον ε, εξωτερικής ανάθεσης, με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι η λιανική τιμή που πληρώνουν οι, οι, τελικοί καταναλωτές. Εδώ με το κίτρινο βλέπετε εκείνες τις δικαιοδοσίες που αναφέρονται στο υπολογισμένο κόστος εξωτερικής ανάθεσης για λιγότερο από ένα ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με το TTF, που είναι δηλαδή ο μέσος όρος για την Ευρώπη. Το γαλάζιο είναι 1 με 3 ευρώ και το σκούρο μπλε είναι πάνω από 3 ευρώ. Και αν δείτε υπάρχει πολύ περισσότερο κίτρινο, το οποίο αναδύεται με το πέρασμα των χρόνων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το κίτρινο επεκτείνεται από το κέντρο και όχι από την περιοχή από την οποία έρχεται το φυσικό αέριο. Δηλαδή, το κόστος της ανάθεσης ε, εξαρτάται περισσότερο από την ανταγωνισμό στις αγορές παρά από την εγκύτητα ή την ε, απόσταση την μεγάλη απόσταση από την προέλευση του φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός είναι θετικός για τον τελικό καταναλωτή. Βλέπουμε λοιπόν πως ήδη έχουν ωφεληθεί, ε, πρόκειται για δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2013, τα οποία τα περισσότερα προκύπτουν, προέρχονται από την αλλαγή στους μηχανισμούς τιμολόγησης των μακροχρόνιων συμβάσεων, όπου όλο ένα και περισσότερο βασίζονται σε τιμές του κόμβου και όχι στις τιμές του πετρελαίου. Και αυτές οι τιμές δηλαδή ωφελούνται από τον ανταγωνισμό στην αγορά. Τώρα, αγορά ηλεκτρισμού. Εδώ βλέπετε τρία γραφήματα. Το ένα είναι πού βρισκόμαστε με την ε, σύνδεση των αγορών. Η περισσότερο τμήμα της Ευρώπης είναι συνδεδεμένο. Από τα στενά του Γιβραλτάρ μέχρι τη θάλασσα Μπάρεντ φτάνουμε και καλύπτονται έτσι ε, πολλές δικαιοδοσίες. Μετά έχουμε κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρουμανία και άλλες χώρες που θα, μπουν, ε, ε, που θα συνδεθούν σύντομα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό ότι έτσι έχουμε μπορέσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούνται οι ε, διασυνοριακές συνδέσεις. Δεξιά βλέπουμε κάτω το επίπεδο απόδοσης. Πώς χρησιμοποιούνται και πού χρησιμοποιούνται σωστά οι δομές όταν υπάρχει διαφορά κόστους. Έχουμε κερδίσει 26% αποδοτικότητα στη διάρκεια αυτής της σχεδόν δεκαετίας. Αυτό όμως δεν είναι εγγυημένο. Εκεί που δεν λειτουργεί η σύνδεση της αγοράς, εκεί πάμε αντίθετα σε αυτή την τάση. Υπάρχει χώρος δηλαδή αν και έχει υπάρξει βελτίωση, υπάρχει χώρος για βελτίωση και εξισορρόπηση των αγορών. Όπως γνωρίζετε, το, η δέσμη για την καθαρή ενέργεια προβλέπει ότι τουλάχιστον το 70% της γενικής ε, δυνατότητας θα πρέπει να διατίθεται για εμπόριο. Αυτό ήταν ζήτημα μέχρι τώρα, γιατί περισσότεροι από την ε, διασυνοριακή δυνατότητα δεν μπορούσε να μπει στην αγορά, διότι δεσμεύεται να λάβει υπόψη την εσωτερική συμφόρηση. Εδώ έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εάν δείτε πού έχουμε το NTC, δηλαδή εκεί όπου μπορούμε να υπολογίσουμε την, ε, τις δυνατότητες και την ε, απόδοση, είμαστε ακόμα κάτω από το, από το επιθυμητόριο. Αν δούμε όμως ε, το άλλο διάγραμμα στα δεξιά, βλέπουμε ότι εκεί επιτυγχάνεται ο στόχος. Ενώ στα αριστερά βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν, γιατί ο νέος στόχος είναι επιχειρησιακός και πρέπει να τηρηθεί ε, την πρώτη πρώτη του επόμενου έτους. Τώρα, ασφάλεια ανεφοδιασμού και η λειτουργία των μηχανισμών ε, κάλυψης που πρέπει να λάβουν υπόψη την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Όμως αυτοί οι μηχανισμοί ε, λειτουργούν ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες ή τουλάχιστον σύμφωνα με την εκτίμηση του, ε, τις μας δεν υπάρχει ανησυχία. Αυτές που καλύπτονται από το κόκκινο είναι αυτές που εφαρμόζουν τους μηχανισμούς αυτούς ακόμα και αν με βάση την εθνική SOE δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα προσαρμογής ούτε το 2020 ούτε για το 2025. Σε ορισμένους από αυτούς τους μηχανισμούς ε, επιβάλλεται το κόστος τους στον καταναλωτή. Και τελική διαφάνεια, να σας δείξω και πάλι τι είδους ωφέλη έχει επιφέρει αυτή η διαδικασία. Στο πράσινο χρώμα Βλέπουμε την αξιολόγηση των ωφελών που έχουν ήδη δοθεί από την ε, σύνδεση των αγορών. Έχουμε ένα δισετησίως, πάνω από ένα δισετησίως. Περισσότερα πρέπει να γίνουν ακόμα για την ε, αγορά και όσον αφορά το πλαίσιο υπολογισμού δυνατοτήτων, που θα επανέλθω σε αυτό στις ερωτήσεις αργότερα, όσον αφορά την ασφάλεια ανεφοδιασμού, αλλά και ενδεχομένως τη δυνατότητα νέου συντονισμού όλων αυτών. Αυτά έχω να σας πω λοιπόν για σήμερα και όπως είπα είναι η τελευταία μου ε, φορά που έρχομαι εδώ για να σας ε, παρουσιάσω την ετήσια έκθεση της ε, αγοράς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας εδώ στην Επιτροπή Ήτρη και για, γενικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το οποίο συνεργαστήκαμε αγαστά πριν ακόμα δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός. Σας ευχαριστώ πολύ και με τα χαρά με τη συνάδελφο Κλάρα Πολέτη να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ξεκινάμε με τους δανειστές. Κυρία Καρβάλ, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση, για το έργο σας, για το χρόνο που αφιερώσατε όλο αυτό το διάστημα και τις καλές σχέσεις που είχατε με την Επιτροπή μας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη λειτουργία της οστρικής αγοράς φυσικού αερίου. Πρώτον, κάποιες από τις διασυνδέσεις καθυστερούν. Δεν σημειώνεται πρόοδος. Υπάρχει μια έκθεση όπου τα παρακολουθείτε αυτά Ποιο πιστεύετε ότι είναι ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό. Αναφέρομαι, παραδείγματο χάρη, ε, στην Ιβυρική, Χερσόνησο, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία. Αυτά τα project ε, δεν προχωράνε. Τι συμβαίνει τελικά. Δεύτερο ερώτημα σχετικά με το φυσικό αέριο. Αυτές οι διασυνδέσεις ε, που ε, μεταφέρουν το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, ε, για πιο καθαρά οχήματα ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφερθήκατε σε δύο καταστάσεις στην Ευρώπη. το, Δύση με τον Νότο και το, που είναι απόλυτα συνδεδεμένα και τα νέα κράτη-μέλη που δεν είναι πια νέα βέβαια ε, που, όπου όμως ακόμα υπάρχουν προβλήματα με την ε, ενιαία αγορά ε, για αυτούς. Πώς βλέπετε το μέλλον για την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελευταίο ερώτημα, σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό δυνατοτήτων, είπατε ότι κάποιες από τις χώρες που έχουν ήδη εφαρμόσει το μηχανισμό αυτόν ε, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, ανεφοδιασμού, ασφάλειας ανεφοδιασμού. Ε, και αυτός είναι ένας λόγος για τους οποίους πληρώνουν περισσότερα οι καταναλωτές. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι βέβαια. Ε, θα πρέπει νομίζω να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον καταναλωτή εδώ, μεγαλύτερη προσοχή, να μην είναι αυτός ο οποίος πλήττεται, κάθε φορά. Βεβαίως και πρέπει να πληρώσει μια δίκαιη τιμή. Όταν ένα κομμάτι έχει να κάνει κλιματική αλλαγή, λογικό είναι να πληρώσει καταναλωτή. Αλλά υπάρχει μια λογική φορολόγηση, ε, φόρου πάνω στου φόρου και επιβαρύνεται πολύ ο καταναλωτή. Στον τομέα τη ενέργεια πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, πιστεύω, ε, στον καταναλωτή και στι ανάγκε του. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι οι συντονιστέ έχουν τρία λεπτά για τις παρεμβάσει τους και τα υπόλοιπα μέλη δύο λεπτά. Για τους ελθές και δημοκράτες, παρακαλώ κυρία Κουταγιάρ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι της έκθεσης που έχει να κάνει με τις τιμές λιανικής για την ηλεκτρική ενέργεια. Από το 2008 και μετά οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά έχουν αυξηθεί κατά 28,4%. Ονομαστική αξία, έτσι. Υπάρχουν κάποιες επιβαρύνσεις, ε, ε, πρόσβαση στο δίκτυο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, είναι η βασική λόγοι αυτή ε, για την αύξηση. Ε, το νέο, η νέα πράσινη συμφωνία, το νέο Green Deal θα προωθήσει ακόμα περισσότερο ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι θετικό. Ποιος θα είναι όμως ο αντίκτυπος ε, στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μέσα εισοδήματα και με περιοχές που οικονομικά δυσκολεύονται. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την συγκεκριμένη πρόκληση, έχετε εντοπίσει κάποιες λύσεις για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση και τα εργαλεία αυτά θα προωθηθούν από το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, ε, θα αρκέσει αυτό το πακέτο, έχετε σκεφτεί κάποιες κρατικές γραμμές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας ε, για να προστατευθεί η αγορά από υπερβολικά ψηλές τιμές και κυρίως πώς ε, βλέπετε το ρόλο σας για την εφαρμογή του νέου Green Deal. Αυτό απευθύνεται κυρίως ε, στον διάδοχο, στη διάδοχό σας. Μάλιστα για τη Renew τώρα ο κύριος Πέτερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή δουλειά σας για να προωθηθεί ε, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντικά τα καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Ήθελα να σας συγχαρώ για όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι έχετε βρει κάποιους λόγους για αισιοδοξία στην πιο πρόσφατη έκθεσή σας για την περαιτέρω ε, ενοποίηση, ολοκλήρωση της αγοράς. Ε, τρία θέματα θέλω να θίξω για το κόστος της μη ολοκλήρωσης. Μας δείξατε, μας δείξατε κάποιες διαφάνειες, μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα ακόμα όμως ε, για να δείξετε στην Επιτροπή μας ε, πόσο σημαντικά είναι τα ωφέλη εάν συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο στενά. Δώστε λίγο έμφαση σε αυτό αν θέλετε. Δεύτερον, υπάρχει πάρα το δημοσιονομικό ζήτημα. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήταν και χρήσιμο για την Επιτροπή μας να μας πείτε εσείς ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον παρόντο προπολογισμό, ε, πώς βλέπετε τις δυνατότητες που έχει η υπηρεσία ε, να παίξει το ρόλο της, να αναλάβει τα καθήκοντά της με βάση τα υπάρχοντα δημοσιονομικά στοιχεία. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα όρια και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε εφόσον παραταθεί ο παρόν προπολογισμό. Πέστε μας λοιπόν και από αυτού κάτι. Και τέλος, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή ξεκινήσει μια συζήτηση, μια αξιολόγηση των PCIs. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας. Είχαμε αυτή τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες ε, και τώρα πάλι ξανά ε, γίνεται αυτή η συζήτηση με διάφορες μορφές. Εσείς πώς το βλέπετε, ε, πώς βλέπετε τους καταλόγους των PCIs, ε, πρέπει να βρεθεί, βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας για να πετύχουμε τους στόχους των Παρισίων για το κλίμα. με βάση τις γνώσεις σας, την πραγματογνωμοσύνη σας, πιστεύετε ότι ακολουθούμε τη σωστή οδό για τα PCIs και αν όχι τι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποτότσινικ και χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ και τώρα για τους πράσινους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ποτότσνικ, λέει ο κύριος Καφ, ε, ήσασταν ε, πολύ αποτελεσματικό στα καθήκοντά σας όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ο κάθε νέος κύκλος ε, όμως φέρνει νέες προκλήσεις. Ε, το ευρωπαϊκό Green Deal είναι μια πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία. Πριν όμως μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό Green Deal, πρέπει να μιλήσουμε για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να αναφερθώ στις επιπτώσεις αυτού. Η υπηρεσία έχει μια σειρά από υποχρεώσεις να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στην αγορά, την παρακολούθηση, την καταπολέμηση της απάτης, ε, ε, την πρόληψη. Ε, όμως τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη πόρων δεν έχει επιτρέψει στην Άκερ να παίξει το ρόλο της πλήρως. Το Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί για τις δραστηριότητές σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και σας έχουμε υποστηρίξει στην προσπάθεια να βρείτε τους, φο, τους πόρους ε, οικονομικούς και ανθρώπινους που χρειάζεστε. Και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σημαντικό ε, εισφορέα στου πόρους αυτούς Από ό,τι φαίνεται όμω οι πόροι αυτοί μετά το Brexit ε, δεν θα υπάρχουν και δεν είναι σαφές ακόμα εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει, ε, ως, θα παραμείνει στο εσωτερικό της αγοράς ενέργειας. Πρόσφατα έγιναν κάποιες συζητήσεις για την υπηρεσία που θα δημιουργήσει τους, τους δικούς της ιδίους πόρους και θα επιβάλλει κάποια τέλη στους συμμετέχοντες στην αγορά για να μπορέσει ε, να παράσχει αυτή την υπηρεσία μιας λειτουργούσας αγοράς. Όμως, πολύ απλά ρωτάω, ποια βήματα θα πρέπει να κάνουμε έτσι να μπορέσει η Aker ε, να συλλέξει αυτά τα χρήματα που συμμετέχοντες στην αγορά ε, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, την διαφάνεια και την ολοκλήρωσή της. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα. Πώς αξιολογείται τον αντίκτυπο του Brexit στην ε, διαφάνεια ε, της αγοράς. Και βεβαίως ε, κάτι παράπλευρο εδώ. Ε, τα αποθέματα, ε, τα αποθεματικά δεδομένων στο Μένο Βασίλειο θα είναι προσβάσιμα σε εσά μετά το Brexit. Ε, γενικότερα ο αντίκτυπος του Brexit ε, στις εργασίες σας ε, ποιος θα είναι. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο από την ID θέλει κάποιος το λόγο, ο κύριος Καπά όχι Τώρα είναι η δική μου πολιτική ομάδα. Εγώ είμαι ο συντονιστή. Οπότε να θέσω εγώ το ερώτημα, λέει ο πρόεδρο. Μου έκανε εντύπωση ε, που κάνετε και μια κάποια κριτική σε ό,τι αφορά τα capacity markets. Ε, αλλά οι αγορέ αυτέ ε, δυνατοτήτων ε, προσπαθούν να αλλάξουν και το ενεργειακό μείγμα, έτσι ε, ποια είναι η δική σας άποψη τελικά γι' αυτό. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη ε, θέσπισης και ανάπτυξης αυτών των capacity markets επειδή μιλάμε για το φυσικό αέριο και εμεί ανησυχούμε για την ασφάλεια ανεφοδιασμού ε, και το μέλλον του φυσικού αερίου η ασφάλεια του ανεφοδιασμού είναι κάτι που συνδέεται και με την εσωτερική αγορά και την εξάρτησή της, τις τρευλώσεις που μπορεί να υπάρξουν εφόσον είναι ένας προμηθευτής, ιδιαίτερα για κάποιες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, ε, αλλά και τη Γερμανία, είναι ένα ζήτημα. Εσείς ε, πώς το βλέπετε αυτό, πώς το αξιολογείτε. Αυτά. Αυτά ήταν τα δύο ερωτήματά μου. Και τώρα, κόβε το μικρόφωνο όμως του Προέδρου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Ο κύριος Μπλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστώ και τον κύριο Ποτότσνικ, λέει η κυρία Πάουλου που μας ενημερώνεται. Θα ήθελα να πω για την ε, διασύνδεση ότι η χρήση διασύνδεση έχει γίνει πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν στοιχεία διασύνδεση που χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο ε, για την ε, εμπορία ηλεκτρική ενέργεια. Όμω, ε, επειδή έχω μιλήσει με τεχνικού στη δική μου χώρα, στη Γερμανία, από ό,τι φαίνεται στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν αυτά τα στοιχεία διασύνδεση για να σταθεροποιήσουν το δίκτυο. Εάν δεν μπορούν να το κάνουν πια αυτό, χρησιμοποιώντα αυτά τα στοιχεία διασύνδεση, θα χρησιμοποιούν ε, κάποια άλλα μέτρα και τελικά το κόστος για τον καταναλωτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι τα μέτρα αυτά θα προσθεθούν, ε, θα προσθέσουν μάλλον ε, κάποια ακόμα τέλη, κάποιες επιβαρύνσεις, οπότε θα αυξηθεί το κόστος για τον καταναλωτή. Δεν μπορεί να πληρώσει τόσα πολλά ο ίδιος ο κλάδος για το δίκτυο, οπότε θα ήθελα να ξέρω πώς το βλέπετε εσείς το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. This was... Ευχαριστώ. Αυτά, αυτή ήταν η κυρία Πάουλος. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μπλος. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημά μου αργότερα. Go to the answers and then once again Floss. is your, I don't know how you divide the work. Yeah, but... Λοιπόν, χωρίς τις απαντήσεις σας, όπως θέλετε απαντήστε με ποιο σειρά θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις με την σειρά με την οποία μου τις θέσατε. Ε, αρχικά όσον αφορά την εσωτερική αγορά αερίου Ρωτήσατε για ποιο λόγο τα προγράμματα δεν ε, προχωρούν. Αναφέρατε ότι παρακολουθούμε την ε, πρόοδο και ε, κάθε χρόνο βρίσκουμε ότι το μισό κομμάτι έχει καθυστερήσει. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ακόμα θεωρούμε ότι η αδειοδότηση είναι ένας από τους τομείς όπου εντοπίζεται καθυστέρηση απαιτείται 3,5, ε, απαιτούνται 3,5 χρόνια για την αδειοδότηση. Σε άλλες τώρα ε, περιπτώσεις υπάρχουν επιφυλάξεις από την πλευρά των εθνικών αρχών όσον αφορά την ε, χρησιμότητα των προγραμμάτων και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου ένα πρόγραμμα ό,τι φαίνεται δεν αυξάνει ε, τις ε, ικανότητες ε, και έτσι λοιπόν με βάση την μεθοδολογία φαίνεται ότι δεν έχει ένα θετικό όφελος. Επίσης έχουμε ένα θέμα όσον αφορά την τρέχουσα μεθοδολογία όσον αφορά το αέριο. Εκεί υπάρχει δυσκολία στο να επιλογίσουμε το ωφέλη και σε πολλές ε, ε, περιπτώσεις ε, δεν παρέχεται το κόστος του προγράμματος και έτσι λοιπόν είναι δύσκολο να έχουμε μια τέτοια ανάλυση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εμποδίζει τα προγράμματα γενικότερα είναι η ε, φάση της αδειοδότησης. Επίσης αναφερθήκατε στο θέμα της ε, ε, τρέχουσας υποδομής, της υπάρχουσας υποδομής για το αέριο που έχει απαλλαγή από εκπομπές αερίου. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά υδρογόνου ή άλλων αερίων. Θα υπάρξει μια φάση μετάβασης όμως ε, κατά τη διάρκεια, τη οποία θα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα χρειαζόμαστε πάνω από ένα δίκτυο, κάτι το οποίο δημιουργεί ε, ανησυχίες όσον αφορά το κόστος ε, και είναι και η, η πρόκληση του να χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο ήδη έχουμε για να μας βοηθήσει στη διαδικασία της ε, απαλλαγής από εκπομπές. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για την Επιτροπή που δεν έχει συσταθεί ακόμα, όμως ε, ε, πιστεύω ότι από όσα ακούω ότι η Επιτροπή σκέφτεται να προτείνει κάτι ε, για το θέμα αυτό ε, το οποίο θα αφορά τον τομέα του φυσικού αερίου. Τώρα στην αγορά ηλεκτρισμού αναφερθήκατε στο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην αγορά δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Στον τομέα του ηλεκτρονισμού δεν έχουμε τόσο έντονο αυτό το χάσμα. Υπάρχουν δύο τομείς ε, που θα πρέπει να συγκληθούν. Όμως ε, αυτή τη στιγμή ε, το, η σύγκληση για τις τέσσερις καφέ χώρες στο χάρτη περιμένουν την εφαρμογή θα ακολουθήσει σύντομα η διαδικασία. Τέλος πάντων. Ορίστε, σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε αυτό τον χάρτη. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν το οποίο να τις αποτρέπει να συγχωνευθούν εφόσον ε, ε, προχωρήσει η διαδικασία στο αέριο η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερη ορίμανση στις ε, ε, δυτικές αγορές, ε, κάτω για παράδειγμα, και η Βρετανική αγορά επίσης. Η Ανατολική αγορά τώρα βασίζεται κυρίως στα καύσιμα. Τώρα οι μηχανισμοί ικανοτήτων εδώ ανησυχούμε ότι επειδή ε, το κόστος είναι αυξημένο, το ε, νέο πακέτο ε, παρουσιάζει διάφορα, διάφορα βήματα μέχρι ότου να εισαχθεί ο νέος ε, μηχανισμός. Ένα από τα βήματα είναι μια ανησυχία που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μέσα της αγοράς και αυτό, αυτή είναι η αξιολόγηση την οποία διεξάγουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε, εξετάζοντας την περίοδο 20 20-25 υπάρχουν ανησυχίες λοιπόν οι οποίες μπορεί να ετυλιγούν την ε, δημιουργία αυτού του μηχανισμού διότι εάν ε, δημιουργηθούν χωρίς κάποια αιτιολόγηση τότε μπορεί να ε, επιβάλλουν επιπρόσθετο κόστος στους καταναλωτές. Τώρα όσον αφορά την, το λιονικό τη λιανική ε, αγορά σχετικά με το ε, ηλεκτρισμό και, την, ε, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες οι οποίες προστίθενται αυτή τη στιγμή ίσως να μην επιβάλλουν επιπρόσθετο κόστος αυτή τη στιγμή. Είναι γενικό αυτό. Οι ανανεώσιμες σε σχέση με τις ανανεώσιμες που εμφανίστηκαν στο παρελθόν βλέπουμε διάφορες εναλλακτικές για παράδειγμα, για ε, την παράδοση ανανεώσιμων με, μηδέν, με μηδενικό επιβρόσθετο κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, εξάλληψη άνθρακα, εκπομπών άνθρακα. Οι νέες ανανεώσιμες δεν πρόκειται να επιβάλλουν το νέο κόστος, νέο κόστος όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση πάνω σε αυτό. Δεν είναι στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας να παράσχει κατευθυντήριες πάνω σε αυτό. Εμείς απλά παρακολουθούμε αφορά περισσότερο τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα υποστηρίξουν αυτά τα ζητήματα. σχετικά με το κόστος της ενσωμάτωσης. Έχω αυτό εδώ το διάγραμμα, το κόκκινο αφορά το κόστος της ε, μη ενσωμάτωσης, έχουμε δηλαδή τα ωφέλη τα οποία θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στους καταναλωτές σε που μπορούσαμε να ε, ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία, ανέφερα ότι έχουμε ε, τη δυνατότητα να απελευθερώσουμε μέχρι και ένα δισεκατομμύριο ε, μέσω της σύζευξης της αγοράς. Υπάρχουν ακόμα κάποια όρια όπου πηγαίνουμε προς τη λάθος κατεύθυνση. και υπάρχουν και άλλοι τομεί όπου θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τον σχεδιασμό της αγοράς. Ε, οι τομεί αυτοί αναφέρονται σε αυτήν εδώ την εικόνα και αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τομείς ε, με ορθό τρόπο, τότε θα μπορέσουμε ε, να παραδώσουμε ωφέλη στους κατανοητές. Ναι, λοιπόν, η διαδικασία ήταν επιτυχημένη, έχει αποφέρει αποτελέσματα και θα ήθελα να αναφέρω ότι ο σχεδιασμός για την αγορά ηλεκτρισμού είναι ο πιο φιλόδοξος ε, παγκοσμίω όσον αφορά την ε, γεωγραφική κάλυψη και τον βαθμό της ενσωμάτωσης της αγοράς. Πολύ συχνά λοιπόν ακούμε αυτούς που τα εξετάσουν αυτά τα θέματα. Ακούμε το PJM για το PJM στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ ε, το PJM εκεί είναι ουσιαστικά η Γερμανία και η Πολωνία μαζί σε εμά. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά, όμως η αγορά μας είναι πολύ πιο φιλόδοξη ε, και ε, αυτά είναι τα ωφέλη τα οποία θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στου καταναλωτέ. Τώρα το ζήτημα του προπολογισμού γνωρίζω ότι ε, σας απασχολεί αυτό μαζί με εμάς και χαιρόμαστε που μας έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό. Υπάρχουν δύο θέματα, από τη μία τα χρήματα, από την άλλη οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή στην ε, περίπτωση ε, του, ε, του πλαισίου μας και την εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς της αγοράς οι συνάδελφοί μου ε, δεν μου δίνουν ε, ακριβείς αριθμούς. Ε, αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε το 20% της αγοράς, δεν λέμε ποιο 20% ακριβώς και αλλάζουμε συνεχώς, όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφαρμόζουμε τον κανονισμό έτσι όπως πρέπει, την εντολή μας όπως πρέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο Υπάρχουν άλλα ε, κόστη τα οποία έχουν αναφερθεί από τις εθνικές, εθνικές διοικήσεις ε, για την επιβολή προστήμων. Νομίζω πέρσι είχαμε ένα πρόστιμο 5 εκατομμύριων. Ε, αυτά είναι οι, ε, αφορούν συμπεριφορές που δεν θέλουμε να βλέπουμε στην αγορά και όταν ε, τις εντοπίζουμε και υπάρχουν κυρώσεις ε, τότε λειτουργούν αποτρεπτικά. Χαίρομαι λοιπόν που ε, για αυτό το κομμάτι της αγοράς το οποίο έχουμε εξετάσει δεν έχουμε βρει άλλες ε, παραβάσεις. Ε, είμαστε καλύτερα από ότι οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Όμως αν δούμε τον κατάλογο των νέων εργασιών που ανατίθενται στην υπηρεσία, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με τους πόρους που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δοκιμάσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, ε, μια λαθασμένη αναλογία όσον αφορά την ε, φιλοδοξία που έχουμε και τα έξοδα. Έχουμε, θέλουμε 40 επιπλέον προσωπικό, άτομα προσωπικό, το κοινοβούλιο ε, μας είπε ότι ε, θα δούμε ε, τι μπορεί να προκύψει από τους τριμερείς διαλόγους. Τέλος, τα PCI και η φιλοδοξία των Παρισίων είναι μια μετάβαση την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε υπάρχουν υποδομές ε, ε, στα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα του φυσικού αερίου ε, και επίσης θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτή είναι η συνολική, η συνολική μας δράση για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της δέσμευσης για την Συμφωνία των Παρισιών. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση για το Brexit, αυτό το οποίο ε, θα συμβεί εξαρτάται από τους όρους με τους οποίους θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σκληρό Brexit ε, και ήδη μας έχει ενημερώσει η Επιτροπή σημαίνει ότι ουσιαστικά ε, θα κλείσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο από τη στιγμή που θα αποχωρήσει. Δεν θα μας βλέπουν, δεν θα τους βλέπουμε. Οπότε θα είναι κάτι ε, ατυχές να συμβεί κάτι τέτοιο, να το πω ε, ε, απλά. Αυτό ιδάλλως, ε, αν υπάρξει συμφωνία, θα παραμείνει στην παρακολούθηση για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας. Όμως δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, διότι δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Κύριε ε, Πρόεδρε, αναφερθήκατε για τις ικανότητες της ε, αγοράς, αναφέρθηκα σε αυτό και επίσης τώρα για την εξάρτηση στο αέριο. Πιστεύω ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Έχουμε βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά την ε, διασύνθεση από το 2009 και την κρίση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράσχει στην Ουκρανία αέριο ρωσικό, όμως από τα δυτικά. Το μοντέλο, μας, το μοντέλο μας σχετικά με τους στόχους ε, για το αέριο έχει συγκεκριμένους ε, στόχους ε, σχετικά με την απόκτηση αερίου, όμως ακόμα υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν μια ε, κληρονομιά όσον αφορά την μία πηγή τη μία προέλευση και ελπίζω λοιπόν ότι ε, μελλοντικά ύστερα από μία πρόταση ε, της Επιτροπής ε, θα εξετάσουμε και το πώς η δυσλειτουργία της αγοράς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί μέσω της νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή για το 2015 είχαμε προτείνει μια σειρά μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθήσουμε και σε περίπτωση που εντοπίσουμε προβλήματα ε, τότε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Δεν έχουμε δει πολλά πάνω σε αυτόν τον τομέα. Είχαμε δει κάποιες συγχωνεύσεις περιοχών ε, που βελτίωσαν την λειτουργία της αγοράς. Παρ' όλα αυτά απαιτείται περαιτέρω δράση πάνω σε αυτό. Και τέλος όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Πάουμς. Έχουμε δύο ζητήματα εδώ. Ε, σε τι βαθμό οι ικανότητε των ε, διασυνδετών ε, χρησιμοποιούνται για τον τομέα αυτό. Έχω, δι, έχω δύο αποτελέσματα πάνω σε αυτά. Ένα, από ότι, ένα αφορούσε την αποτελεσματική χρήση των όσων έχουμε και δεύτερον το τι ε, μας διατίθεται. Υπάρχει μια ισορροπία βλέπουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για το εμπόριο το οποίο έχει τα ωφέλη του Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ποια είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ του εμπορίου και της ε, χρήσης για άλλους ε, σκοπούς. Ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή και το Συμβούλιο μάλλον αποφάσισαν για την ισορροπία στο 70% και εμείς παρακολουθούμε εάν αυτό θα επιτευχθεί, πότε και πώς αυτή τη στιγμή όμως ε, με τα βεβαιότητας, ε, κάτι το οποίο το έχει τονίσει και εδώ και χρόνια η υπηρεσία, είναι ότι η διαθέση για εμπόριο είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι θα μπορούσε, ε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί ο κ. Διευθυντή ε, απάντησε εκτεταμένα σε όλε τι ερωτήσει. Εγώ ήθελα απλά να αναφερθώ σε μια ερώτηση που αφορούσε το ρόλο του ΆΣΕΡ στην ε, εφαρμογή τη νέα πράσινη συμφωνία. Ο ρόλος του Άσερ θα είναι κρίσιμος, γιατί είναι ένας οργανισμός για τη συνεργασία ανάμεσα στου ρυθμιστέ ενέργεια. Αυτέ οι συγκριτικέ προσεγγίσεις θα είναι ακόμα πιο σημαντικέ για το μέλλον, γιατί θα ε, χρειαστεί να αλλάξουμε πραγματικά και να επιταχύνουμε την αλλαγή στα ενεργειακά μας συστήματα, <clears throat> αλλαγή που πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε αρκετά ευέλικτες λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε να καλύψουμε μάλλον τις εθνικές ανάγκες, αλλά να είναι και αρκετά εναρμονισμένος ώστε η αγορά να λειτουργεί ε, αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας συντονισμός ανάμεσα στην ευρωπαϊκή άποψη και την εθνική άποψη και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια, να δούμε δηλαδή τη λειτουργία των αγορών μέσα σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Τώρα πρέπει να δούμε το μακροπρόθεσμα μηνύματα προς την αγορά ώστε να γίνει η μετάβαση και Μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι υπάρχει μέγας ρόλος για την ανάπτυξη υποδομών, το συντονισμό ανάμεσα στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, το νέο είδος ενέργειας, τα νέα είδη μάλλον ενέργειας, γιατί χρειάζεται συντονισμένη εικόνα για όλες τις υποδομές ενέργειας, λειτουργία της αγοράς και καλύτερη ολοκλήρωση ανάμεσα στις ε, ε, διάφορους φορείς ενέργειας. Αυτή η ολιστική προσέγγιση θα είναι πολύ, πολύ κρίσιμη. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, σας ευχαριστήσω και του Ποτόσκι για την εξαιρετική σας εργασία. Εννέα χρόνια ήσασταν σε αυτή τη θέση. Μάλιστα. Mm. Ωραία, λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η συζήτηση με τον υποψήφιο διευθυντή του ΑΣΕΡ, κύριο, του Άσερ, κύριο Τσίγκλερσεν. Ε, ο κύριος Κρίστιαν Σίγγελσεν είναι ο υποψήφιος διευθυντής ε, του ΆΣΕΡ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει τον κύριο Τζίγκλερσεν ως νέο διευθυντή του οργανισμού για μια θητεία πενταετίας που ξεκινά την 1η Πρώτου του 20, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού περί ΑΣΕΡ 2019 942 ο κύριος Τσίγκλερσεν θα κάνει τη δήλωσή του και μετά θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτή την παρουσίαση. Και πάλι έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας για αυτό το ε, θέμα. Έχετε το λόγο κύριε Τσίγκλερσεν. Για την αρχική σας εισήγηση έχετε 10 λεπτά και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Very uh, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να σας πω ότι προσέβλεπα σε αυτή τη στιγμή εδώ και αρκετό καιρό. Ξέρω πως ε, υπάρχει μεγάλη προσήλωση στην, ολοκλήρωση, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Ενέργειας και από τη δική σας Επιτροπή, αλλά και το ίδιο και για το ρόλο του Άσερ σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Για μένα είναι επιστροφή ε, στα πάτρια, ε, γιατί πριν από 15 χρόνια δούλευα εδώ στις Βρυξέλλες και κάλυπτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περνούσα αρκετό χρόνο εδώ στην Ήτρε και πίσω-πίσω, στα πίσω-πίσω καθίσματα παρακολουθούσα τις εργασίες και είναι, αισθάνομαι ευχάριστα που βρίσκομαι πάλι εδώ, αν και θα έχω τώρα διαφορετικά καθήκοντα τελώς. Ε, να σας πω λοιπόν σύντομα ποιο είναι το δικό μου όραμα για το Άσερ, δεύτερον ποια είναι τα... Ε, ποιοι θα είναι οι στόχοι, οι άμεση αλλά και οι μεσοπρόθεσμοι, ε, τις βασικές αλλαγές που θα περάσει η αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και τι θα σημάνουν από οργανωτικής άποψης αυτές οι αλλαγές για το ΆΣΕΡ. Καταρχάς, όπως είδαμε και από την προηγούμενη συζήτηση, τώρα ολοκληρώθηκε. Νομίζω πως ο ρόλος του Άσερ είναι σημαντικός όσον αφορά την αυξημένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην ενέργεια. Και θα σας πω το εξής. Νομίζω πως έχει ρόλο κλειδί να παίξει στο να οικοδομήσει την πίστη στην αυξημένη αμοιβαία εξάρτηση σε αντίθεση με το να μην έχουμε αμοιβαία εξάρτηση και εμπιστοσύνη ε, και να αναζητούμε διαφορετικές λύσεις. Ο Άσερ έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ και συμφωνώ με αυτούς που θεωρούν ω αυξημένο το ρόλο του Άσερ για το μέλλον. Και αυτό γιατί η πάυση χρήση του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ακολουθεί αυξητική τροχιά και θα ήταν ε, νομίζω ένας τρόπος για να ε, πετύχουμε αυτές τις ε, λύσεις με λιγότερο κόστος μέσω της αύξησης των ενεργειακών, της ολοκλήρωσης των ενεργειακών συστημάτων της Ευρώπης. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει κανείς να έχει την πίστη πως θα δουλέψει το σύστημα. Η οικοδόμηση λοιπόν πίστης και αυξημένη αμοιβαία εμπιστοσύνη και εξάρτηση, στο οποίο ο Άσερ θα έχει να παίξει ρόλο κλειδί. Ο, το Άσερ λοιπόν θα έχει να αντιμετωπίσει διάφορα διάφορα έργα στα επόμενα χρόνια όπου θα, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την πίστη. Για τον ηλεκτρισμό, όπως είπε και ο Αλμπέρτο, υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν περισσότερο οι κωδικοί των δικτύων, να υπάρξουν περισσότερες διασυνδέσεις ανάμεσα στις χώρες, να περιφερειοποιηθεί περισσότερο η διευκόλυνση της αγοράς και οι προσπάθειες ε, προγραμματισμού και σχεδιασμού των περιφερειών περιφερειακών φορέων, καθώς και το να έχουμε περιφερειακό πεδίο εφαρμογής που θα προέρχεται όμως από το κέντρο. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει πολύ όσον αφορά την ε, ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια γενική μείωση τη συζήτηση του φυσικού αερίου και αυτό θα επιφέρει κάποια αριθμιστικά ζητήματα όσον αφορά ας πούμε τις τιμές εφόσον έχουμε χαμηλή χρήση ενός μεγάλου δικτύου αυτό έχει επιφέρει θέματα τιμών αλλά και ίσως και θέματα κλεισίματος κάποιων ε, εργοστασίων παραγωγής ε, Μπορεί να τεθούν και θέματα ιδιοκτησίας, αποδέσμευσης και αποσύνδεσης στην πορεία. Επίσης, τα project ε, ηλεκτρισμού θα χρηματοδοτούνται περισσότερο από το PCI, περισσότερο από ό,τι υποδομές για φυσικό αέριο, αν και θα υπάρχουν κάποια προγράμματα για το φυσικό αέριο, στο βαθμό που αυτά θα συντεριάζουν με την πάυση της χρήσης του άνθρακα. Το PCI θα πρέπει περισσότερο να δει τις προσπάθειες διανομής, γιατί πολλές αλλαγές θα γίνουν και στο επίπεδο της διανομής. Και τέλος, για την εποπτεία της αγοράς, τη διαφάνεια και το ζήτημα της εντολής ε, που συζητήθηκε στην προηγούμενη συζήτηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα κάνουμε σωστά, να παραμείνει η εμπιστοσύνη στις ολοκληρωμένες αγορές και ε, ε, ίσως επειδή θα είναι μεγαλύτερες και ανταγωνιστικότερες οι αγορές, θα είναι πιο δύσκολο κανείς να ασκήσει και να βρεθεί σε κυρίαρχη θέση αλλά και η ανείχνευση της ε, εξουσίας στην αγορά θα είναι πιο δύσκολη ακριβώς επειδή θα είναι πιο περίπλοκο το σύστημα. Και έχω ακούσει από συναδέλφους στον Άσυρο ότι καταγράφονται περίπου 3 εκατομμύρια την ημέρα. Άρα λοιπόν το να έχουμε μια κατάλληλη βάση εποπτείας για να το χειριστούμε αυτό θα είναι πολύ βασικό. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά επαρκείς πόρους ώστε να γίνει αυτό αποτελεσματικά. Τώρα, επειδή το Άσερ θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά πρέπει να τα χειριστούμε σε καιρούς ε, ε, ε, ρηξικέλευθων αλλαγών. Όλοι οι τομείς ε, της οικονομίας αντιμετωπίζουν ψηφιοποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και στο ενεργειακό τομέα. Αλλάζουν τα ενεργειακά συστήματα, τα οποία θα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένα στο μέλλον. Η πάυση της χρήσης του άνθρακα επίσης είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και ευκαιρία ταυτόχρονα. Και μάλιστα τα ενεργειακά συστήματα μάλλον θα είναι πιο αποκεντρωμένα στο μέλλον. Βλέποντας λοιπόν όλες αυτές τις αλλαγές που οφείλονται στην άφηση της χρήσης, το Άσερ μαζί με τους ρυθμιστές των χωρών μελών, καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί θα πρέπει να αξιολογήσουν τις προσεγγίσεις τους υπό το φως αυτών των αλλαγών και θα πρέπει να είναι έτοιμο να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν ισορροπία σε δύο βασικά ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς θα πρέπει να εξισορροπηθεί ο ρόλος της πανεπιρωτικής αγοράς που θα είναι πολύ αποτελεσματική και ολοκληρωμένη με αυξημένες τοπικές, τοπικούς μεγάλους κόμβους, ε, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα τα εξορροπήσουμε αυτά τα δύο δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχει κανείς μια κρυστάλλινη σφαίρα να μου πει το μέλλον. Ε, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να βρεθεί αυτή η ισορροπία και θα πρέπει να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το θέμα. Έπειτα επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Πολέτη στα τέλος της προηγούμενης ε, ε, παρέμβασης. Νομίζω πως θα πρέπει να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στο ρόλο των αγορών των αποτελεσματικών αγορών και το ρόλο του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της, ε, του συντονισμού των αγορών ε, σε ένα πλαίσιο ταχεία ταχείας παύσης της χρήσης του άνθρακα. Πρέπει να βρεθεί και μια ισορροπία. Και πάλι δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω με τι θα μοιάζει αυτή η ισορροπία σε 15 χρόνια, αλλά σίγουρα θα μας δώσει δουλειά. Προς τα τέλη λοιπόν το να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημαντικά ε, καθήκοντα και υπό το φως αυτών των σημαντικών αλλαγών στα συστήματα ενέργειας σημαίνει αυτό πως θα έχουμε κάποιες οργανωτικές αλλαγές στο ΆΣΕΡ ε, οι οποίες θα μας, απασχολήσουν από την πρώτη πρώτη που θα αναλάβω καθήκοντα Πρώτη θα είναι ε, να εξασφαλίσουμε μια συνεργασία με τον Άσερ, μια τέτοια προσέγγιση, σίγουρα με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αλλά και με ε, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ε, έπειτα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές, να έχουμε μια προσέγγιση στραμμένη προς το μέλλον, γιατί τα συστήματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και άρα θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές αυτές. Ε, δεύτερον, ε, συμμετοχή των ε, ενδιαφερόμενων φορέων που θα πρέπει να μπορούν να μεταφράσουν τα τεχνικά ζητήματα σε πολιτικές αποφάσεις, πράγμα που κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και έτσι να συμβάλλουμε στη συζήτηση για πολλά από αυτά τα ζητήματα και έπειτα έχουμε και το θέμα των πόρων με τις αλλαγές που γίνονται στα ενεργειακά συστήματα της Ευρώπης, το να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε αρχικά, όπου πιθανότατα θα υπάρχει μεγάλο πριμ για αποτελεσματικές λύσεις και για μεγαλύτερη ολοκλήρωση, πιστεύω πως εκεί θα πρέπει να βρεθούν και οι πόροι που θα στηρίξουν τον Άσερ. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα κλείσω λέγοντας πόσο εκτιμώ την Επιτροπή Ήτρε, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να είναι ενήμερο, να παγρυπνά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Αν με επιτρέπετε επίσης, Πρόεδρε, να κλείσω και 24 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο χρόνος μου και σύντομα να ευχαριστήσω τον κύριο Ποτόσνικ για τις σπουδαίες του προσπάθειες για το ΆΙΣΕΡ, αλλά και για την προσήλωσή του, την δέσμευσή του εδώ, την επαφή του με το Ευρωκοινοβούλιο, γι' αυτό και άλλα θέματα. Ελπίζω λοιπόν πως θα μπορέσω να τιμήσω αυτή το, το, το κληροδότημα συνεργασίας που μου αφήνει. Και προσβλέπω στο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης ε, εκπροσώπους εδώ επισκέπτες. Είναι επισκέπτης της Γιάς Καρβάλιο την Πορτογαλία. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Ήτρε. Και τώρα να ξεκινήσουμε με την κυρία Καρβάλιο από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκερτσεν. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη θητεία σας, τα καθήκοντά σας. Αναφερθήκατε εσείς ο ίδιος στις προκλήσεις και είναι πολλές αυτές που σας περιμένουν. Παρακολούθηση της αγοράς, δημιουργία εμπιστοσύνης, ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού, ψηφιοποίηση, ο συνδυασμός ε, όλων των βασικών στόχων της υπηρεσίας με τις νέες προκλήσεις ε, της απατρακοποίησης ε, θα είναι δύσκολα τα καθήκοντα που έχετε να λάβει αλλά η αποστολή σας είναι σημαντική και όπως πολύ σωστά είπατε δεν υπάρχει ακόμα κάποια τεχνική λύση πλήρη. Πρέπει να συνδυάσουμε ε, την ισορροπία της, στο σύνολο της Υπήρου αλλά και την ευελιξία σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το πακέτο για την καθαρή ενέργεια έχει δώσει μεγάλες ε, δυνατότητες ε, στους καταναλωτές ένας καταναλωτής μπορεί να παράγει ο ίδιος την ενέργειά του, μπορεί και να την πωλεί, δημιουργούνται κοινότητε ενέργεια και αυτό σε ορισμένε περιπτώσεις ε, μπορεί να είναι μια πολύ καλή λύση σε κάποιες περιοχές. Όχι μόνο σε αστικό περιβάλλον, αλλά σε βιομηχανικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα, μπορούμε να έχουμε καλύτερες και πιο καθαρές λύσεις, ε, πιο αποκεντρωμένα και αυτή η εξουσία που δίνουμε στους καταναλωτές ε, έχει αυτό κάτι το συμβολικό. Βάζουμε τους ανθρώπους στο κέντρο των πολιτικών μας. Είναι γενικότερα δηλαδή ε, δίνουμε ε, εξουσίες στους πολίτες. Αυτό είναι κάτι καινούριο στο ενεργειακό πακέτο, αλλά θα είναι σημαντικό αυτό να γίνει σωστά. Και η τεχνική πτυχή δεν είναι απλή οι ρυθμιστικές αρχές ε, είναι αυτές που θα φτιάξουν το interface μεταξύ των δύο λύσεων. Πρέπει αυτό να γίνει σωστά και να δημιουργεί εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές ότι δεν θα υπάρξουν δηλαδή προβλήματα στο σύστημα και διακοπές μπορούν και οι δύο πλευρέ να προχωρήσουν σε ένα κλίμα εμπιστοσύνη χωρί ε, προβλήματα για το σύστημα. Ε, Πολλέ λοιπόν οι νέε προκλήσει, λίγοι όμω οι πόροι, οι ανθρώπινοι πόροι μεταξύ άλλων. Πώ προβλέπετε εσεί ε, να διαχειριστείτε αυτή την υπηρεσία με τον μειωμένο αριθμό προσωπικού και με τόσο σημαντικά καθήκοντα που έχετε αναλάβει για να έχουμε ασφαλή, καθαρή ενέργεια για όλους που είναι αυτό που θέλουμε όλοι στην Ευρώπη και βεβαίως ε, ε, προσβάσιμη οικονομικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουτάγια έχει το λόγο και πάλι για τους S&D. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το έργο σας, το προηγούμενο έργο και το έργο που σας περιμένει. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή Ήτρε. Θέλω να επαναλάβω ένα ερώτημα που έθεσα ε, και στον, στην προηγούμενη ε, πρόεδρο. Μιλούσαμε για το λόγο του Acer ό,τι φορά την εφαρμογή της πράσινη ε, πράσινης συμφωνίας, του Green New Deal. Σίγουρα το Acer μπορεί να συνεχίσει σημαντικά, να βοηθήσει σημαντικά στο ό,τι φορά τον συντονισμό μεταξύ των ρυθμιστικών ταχών, θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά θα ήθελα να έχω και την προσωπική σας άποψη. Πώς σκοπεύετε εσείς να διευκολύνετε αυτό το συντονισμό σε επίπεδο Acer ε, για το νέο αυτό Green Deal. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για την Renew ο κύριος Πέτερσον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ κύριε Τσίγκλερσεν ε, για την θέση αυτή την οποία αναλάβατε. Έχουμε πολλές προσδοκίες. Ε, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Η προκατοχή σας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ε, θέλω να σας ενθαρρύνω να συνεργαστείτε με την Επιτροπή μας όσο περισσότερο γίνεται, διότι μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτή η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά μπορεί να είναι ο πιο καλός σας φίλος. Ε, εμείς ε, πάντως αναμένουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Θέλω να σας ενθαρρύνω απλά να έχετε μια όσο γίνεται πιο στενή συνεργασία με την Επιτροπή μας ε, όπως πολύ καλά, πολύ ορθά έκανε ο προκατοχό σα. Μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η υπηρεσία, έτσι να έρθουν πιο κοντά οι χώρε μεταξύ του ε, και να ε, μοιραστούν τα ωφέλη, όπω φάνηκε από αυτή την έκθεση ε, για την αγορά. Ε, είναι πολλά ακόμα τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να δρέψουμε ε, για τους πολίτες, τους καταναλωτές. Ο ρόλος της υπηρεσίας είναι πολύ σημαντικός γι' αυτό να δοθεί δηλαδή μεγαλύτερη όθηση στην ολοκλήρωση της αγοράς. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός ρόλος εδώ της Acer ως, και ως σύμβουλος, ως ανεξάρτητος σύμβουλος και πολύ σωστά προσπαθήσατε να μεταφράσετε αυτά τα δύσκολα, τα περίπλοκα ζητήματα ε, προς το Κοινοβούλιο αλλά και προς το ευρύ κοινό. Καλώς ήρθατε και αναμένουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα κύριος Μπλος για τους πράσινους. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για αυτή την θέση, για το διορισμό σας. Είναι πολύ σημαντικό, ε, σημαντικός ρόλος σας. Πρέπει να πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση. Ε, έχω να θέσω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα για τα ανοιχτά δεδομένα, την άδεια ανοιχτών δεδομένων ε, στον κανονισμό για την διαφανία. Λέγεται ότι τα, τα δεδομένα για τις, τα, τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού ενέργειας πρέπει να είναι ελεύθερα και προσβάσιμα, όμως σημαντικά δεδομένα όπως ε, οι τιμές παραδείγματος χάρη λιανικής ε, ε, πρέπει να πολιθούν από τις επιχειρήσεις. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες για τους νέους παίκτες στην αγορά. τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα, αλλά όχι με ανοιχτό, με ανοιχτό με ανοιχτή άδεια. το γνωρίζετε το ζήτημα αυτό αναγνωρίζετε ότι το θέμα αυτό δημιουργεί προβλήματα και εμπόδια για νέους παίκτες στην αγορά και τι σκοπεύετε να κάνετε για να απαλληθούν αυτά τα εμπόδια έτσι ώστε να υπάρξει απόλυτη ε, συμμόρφωση με την ανάγκη πλήρους και ελεύθερης ε, πρόσβασης στα δεδομένα. Και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω λίγο προσωπικά να μου πείτε, διότι μίλησατε για την υπηρεσία μεταξύ του ρόλου ε, ε, των, ε, της υπηρετικής, τη της αγοράς Υπήρου και των, τοπικών πρωτοβουλειών, ε, των υποδομών. θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνει εδώ. Επίσης αναφερθήκατε για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και την κατάργηση κάποιων ε, υποδομών. Εδώ μας υπάρχουν νέα project. Πιστεύετε ότι αυτό έχει νόημα, όταν υπάρχει ένα project φυσικό αέριο. Ναι, ευχαριστώ από την IND δεν υπάρχει κάποιος και για το ΕΛΚ θα ρωτήσω εγώ ο συντονιστής και όχι ως πρόεδρος, ο συντονιστής της πολιτικής μου ομάδας. ένα ερώτημα σχετικά με την ε, φτώχεια και τις τιμές. Ε, ο κ. Ποτόλτσνικ νωρίτερα ήταν αισιόδοξο. Είπε ότι αν αναπτύξουμε τις ανώσεις πηγές ενέργειας ε, δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Όμως, αν δούμε τι, τι αναφέρει η δική σας έκθεση, διαπιστώνουμε ότι από το 2008 οι τιμές της, πώλησης, ε, λιανικής πώλησης. Έχουν αυξηθεί κατά 28% από το 2009 μέχρι σήμερα. Ε, υπάρχουν και δεδομένα που μας δείχνουν ότι στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, έχουμε 35% των οικοκυριών που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ε, της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει για 30% των νοικοκυριών στη Βουλγαρία. Οι πολιτικοί μας στόχοι λοιπόν μήπως απομακρύνονται, αποκλίνονται και περισσότερο από την κοινωνική πραγματικότητα σε κάποιες χώρες αλλά βεβαίως ε, αυτό ισχύει και 14% των Ιταλών, 10% των Ισπανών. Ε, θα ήθελα λοιπόν να το σχολιάσετε αυτό παρακαλώ. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα και στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Πίπε από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την ε, νέα σας θέση. Εάν ε, εφόσον ήσασταν σε αυτήν την επιτροπή, τότε γνωρίζετε ότι εμείς προσπαθούμε το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το διαφημίσουμε και στις περιφερειές μας, στους πολίτες. Ε, το έργο μας είναι πολύ θεωρητικό, έτσι ε, λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να πάω ε, και να πω ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Acer. Θα μπορούσατε όμως ε, να μας ε, περιγράψετε το πού θα βρίσκεται η υπηρεσία σε 10 χρόνια και ποια ακριβώς ε, προστιθέμενη αξία συνδέεται με την στρατηγική της Acer, τι θέλετε στα επόμενα χρόνια να επιτύχετε με την συγκεκριμένη υπηρεσία και τι απαιτείται από πολιτικής άποψης ε, και αν το εξηγήσετε έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να το ε, παρουσιάσουμε και εμείς στις περιφέρειές μας τότε πραγματικά θα ενθουσιαστούμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετώντα τον κύριο Ζίγκελσερ και να τον ευχαριστήσω για την εισήγησή του, καθώς και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ε, θέση του αυτή. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι επίγουσα η κατάσταση. Μάλιστα, η υποψήφια πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι οι 100 πρώτες μέρες είναι απαραίτητες για να ε, ευθυγραμμιστεί τη νέα πράσινη συμφωνία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια είναι η δομή του προγράμματος, ε, αλλά για κάτι είμαι βέβαιος, ότι ο ρόλος του ρυθμιστή και συγκεκριμένα ο ρόλος του Ευρωπαίου ε, ρυθμιστή θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικός ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία στις πρακτικές, να εξασφαλιστεί ο έλεγχος ε, του αντικτύπου στις τιμές. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άσερ, ξέρω πόσο καταπληκτική δουλειά κάνατε, πόσο σημαντική είναι ο ρόλος του Ρεμίτ ε, και οι πληροφορίες που μας δίνει και γι' αυτό και θεωρώ πως αυτή η συμφωνία για την αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και της ανταγωνιστικότητάς μας θα δημιουργήσει και κάποιες ε, ε, αλλαγές ε, που θα επιφέρουν ρήξεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην επιτρέψουμε αυτές οι μεγάλες αλλαγές να ορίσουν τη λειτουργία της αγοράς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνο εδώ ένα ταμείο για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ή να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για ειδικευμένους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο, να είναι μια βάση για να ε, βρεθούν νέα μοντέλα στην ε, καινοτομία, στην κατάρτιση, στα πιλωτικά έργα, να δοθεί έτσι μια καθοριστική συμβολή. Εσείς πώς βλέπετε το ρόλο του, του Ταμείου Δίκαιας Μετάβασης μέσα στο πλαίσιο της Πράσινης ε, Συμφωνίας και εσείς πού τοποθετήσετε μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Thank you, thank you. And the next speaker... Ευχαριστώ. Και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος, ε, η κυρία Ράις. Ένα ερώτημα όσον αφορά την εφαρμογή η ενιαία ώρα λειτουργεί σε γενικέ γραμμέ καλά, το οποίο σημαίνει ότι ο ανταγωνισμό ε, σημαίνει υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων και χαμηλότερε ε, τιμέ. Αυτή είναι η όλη ιδέα της εσωτερική αγορά και ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω ύπαρξής της. Όμως όσον αφορά την ενέργεια, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν την πρόσκληση του να αγοράσουν με υψηλότερη τιμή την ενέργεια από ό,τι θα μπορούσε να εισαχθεί με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν να πληρώσουν ε, υψηλότερους λογαριασμούς από ό,τι θα μπορούσαν και παρόλο που υπάρχει η ε, στρατηγική και η σκοπή της ενεργειακής ένωσης. Έτσι λοιπόν ε, με βάση την αρμοδιότητα της Acer πώς ε, θα διασφαλίσετε την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας και ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η κυρία Παύλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Έχω τώρα μια ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της Acer και των νομοθετών όσον αφορά τις διαμάχες ή τις διαφωνίες, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των κρατών μελών. Ε, είμαι από την Γερμανία, οπότε θα καταλαβαίνετε ε, γιατί θέτω αυτό το ερώτημα λόγω του ε, Nord Stream 2, το οποίο είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος ο κύριος Φούλσαν αναφερθήκατε ε, στις ε, μεγάλες αλλαγές που, ε, λαμβάνουν, που συμβαίνουν αυτές τις, τα τελευταία χρόνια. Είπατε ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τις... ανέφερε η κυρία Φοντελάιον ότι θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου υπάρχουν πολλά μέλη τα οποία αγωνίζονται ούτως ώστε το ε, ποσοστό μείωσης να είναι στο 55%. Ε, γνωρίζουμε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ενσωμάτωση της ενέργειας για να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν δηλαδή έχουμε πλεόνασμα ή όταν έχουμε έλλειμμα σε άλλες περιοχές θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή τι πιστεύετε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε πόση ενσωμάτωση χρειάζεται, χρειαζόμαστε και βρισκόμαστε στη σωστή πορεία, ούτω ώστε να επιτύχουμε του στόχου για του οποίου μιλάει η κυρία Φοντελάιαν τη τάξη του 50-55%. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε, θα μπορούσατε να μα δώσετε κάποιε συμβουλέ. Ε, και το δεύτερο ερώτημα είναι, συμφωνούμε όλοι ότι η ενσωμάτωση τη ενέργεια ε, και η εσωτερική αγορά για την ενέργεια είναι κάτι το καλό όταν ε, μιλάμε για γενικού όρου. Όμω έχουμε πολλά προβλήματα ε, όταν ε, θέλουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα κάποιες χώρες μπορεί να μην θέλουν να κάνουν τις επενδύσεις ε, που απαιτούνται οι άλλες περιοχές δεν θέλουν υπερβολική ενσωμάτωση διότι έχουν ανησυχίες σε επίπεδο προστατευτισμού. Πώς λοιπόν αντιλαμβάνεστε το δικό σας ε, ρόλο, πώς ε, μπορείτε να βοηθήσετε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές ε, τις εθνικές επιφυλάξεις. Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχετε και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθηθούμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κύριε Ζίγκλερστεν έχετε τον λόγο. Έρχεται αρκετό χρόνο για να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολλές ερωτήσεις, αρκετές εκ των οποίων θα μπορούσα να πω ήταν, ε, είναι μια πρόκληση. Θα προσπαθήσω όμως να τις απαντήσω όλους, όλες. Ε, θα ε, προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά που ε, τις θέσατε. Κάποιες θα τις ε, απαντήσω από κοινού με άλλες. Κύριε Καβαλιού, μιλήσατε αρχικά για την δυνάμωση των καταναλωτών, για την περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων Ε, θα μπορέσουμε ε, μέσω αυτής της ενίσχυσης να έχουμε την απαραίτητη καινοτομία η οποία θα γίνεται με χαμηλότερο κόστος ε, και φυσικά χρειάζεται και ρυθμιστική καινοτομία ούτως ώστε να ανταποκριθούμε με την ε, καινοτομία στον τομέα της ε, τεχνολογίας και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποσχολήσει τις συζητήσεις μας στην Acer να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και ταυτόχρονα να έχουμε και την απαραίτητη ρυθμιστική καινοτομία ούτως ώστε να υποστηρίξουμε αυτές τις εξελίξεις. Επίσης με ρωτήσατε ε, σχετικά με το θέμα του μειωμένου προσωπικού. Ε, σίγουρα δεν έχω εγκαταλείψει ε, τις προσπάθειες σχετικά με το να έχουμε προσωπικό το οποίο να αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις μας βέβαια φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις, να λειτουργήσουμε με τις όχι άριστα, άριστες συνθήκες Για μένα λοιπόν είναι το τι ε, θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή και το τι ε, μπορεί να ε, δημιουργήσει πίστη για την αμοιβαία υποστήριξη. Αυτοί οι δύο τομείς λοιπόν είναι που θα αποτελέσουν μεγάλη προτεραιότητα για μένα και θα δω πως μπορώ να αντιμετωπίσω ε, και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν τις όμοιες συνέπειες. Ε, αυτό σε, μια, ε, σε συνθήκες όπου θα πρέπει να θέσω συγκεκριμένες προτεραιότητες. Η επιθυμία μου λοιπόν θα είναι να έχω ένα προσωπικό το οποίο να ανταποκρίνεται στο έργο το οποίο μας έχει ανατεθεί. για τους σοσιαλδημοκράτες σχετικά με την Πράσινη Νέα Συμφωνία, ε, θα ε, συνδυάσω και την ερώτηση του κυρίου Φούλσαν. Ε, φυσικά και δεν έχει εκδοθεί ακόμα, όμως δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένος, όμως όσον αφορά τις ε, δράσεις ε, που θα αφορούν και την γενικότερη οικονομία. Σίγουρα θα έχουμε την ε, εξάλληψη των εκπομπών άνθρακα στον τομέα της ενέργειας. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί το μείγμα του ηλεκτρισμού. Είναι επίσης ένα θέμα το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πιστεύω ότι κατά τα επόμενα 10-15 χρόνια θα είναι δύσκολο να δούμε το μονοπάτι το οποίο ε, είναι πιο ξεκάθαρο σε άλλους ε, τομείς όσον αφορά την εξάλληψη των εκπομπών ε, άνθρακα όμως δεν νομίζω ότι ο ηλεκτρισμός θα είναι η μόνη λύση. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τα ενεργειακά συστήματα, πόσο, θα, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η πολιτική ή η τεχνολογία ε, θα πρέπει από ψηφιακή άποψη ε, να ε, η ψηφιακή τεχνολογία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την εξέβριση λύσεων. Ρωτήσατε επίσης το πόσο μπορούμε και σε προσωπικό επίπεδο να τα αντιμετωπίσουμε αυτά από τη στιγμή που θα αναλάβω τη θέση μου στην Acer. Είπα ότι θα πρέπει να ε, κοιτούμε προς το μέλλον, να είμαστε ανοιχτοί προς τις ε, νέες εξελίξεις και θα πρέπει ε, να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας απασχολήσει όσον αφορά την επιφή μας με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές και επίσης πιστεύω ότι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές και τα κράτη-μέλη βλέπουν ε, την κατάστασή τους ε, και θα πρέπει να είναι ανοιχτή όσον αφορά την εξέβρεση ε, λύσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει προτεραιότητα για μένα. Κύριε Πέτιασιν, είπατε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την στενή σχέση της Acer με την Επιτροπή εδώ και θα χαρώ να το κάνω αυτό και θα χαρώ να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε περαιτέρω αυτό με πιο ακριβώς τρόπο από τους ε, πράσινους ε, είχατε αρκετές ερωτήσεις αρχικά όσον αφορά τα δεδομένα. Από ό,τι ε, γνωρίζω θα ήθελα να κάνω μια διαφοροποίηση μεταξύ δύο διαφορετικών στοιχείων από τη μία φορά την διάθεση δεδομέ... από τη μία πλευρά την διάθεση δεδομένων σε data hubs ε, όπου ε, διατίθενται τα δεδομένα στους παράγοντες της αγοράς για να δράσουν με βάση αυτό το οποίο απαιτεί τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των δεδομένων. Πιστεύω ότι αυτό λειτουργεί καλά σε διάφορες χώρες και θα ήθελα να το ε, διαφοροποιήσει αυτό από τα δεδομένα παρακολούθηση, τα οποία είναι απόρριτα πολύ συχνά και ταυτοποιούν κατάχρηση της αγοράς, περιπτώσεις τέτοιες Τώρα σχετικά με το πώς ε, θα μπορούν να γίνουν αυτά τα διαθέσιμα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι απόρριτα, ε, οπότε η απάντησή μου είναι αυτή. Ε, όμως ε, θα μπορούσα να μπω και σε λεπτομέρειες, αν θέλετε άλλες πληροφορίες. Τώρα, το πώς θα υπάρξουν ισορροπίες πάνω σε αυτό, όμως δεδομένου του πώς το πιστεύω εγώ θα πρέπει να υπάρχει ε, μια ισορροπία σχετικά με τον ε, ε, αγορών που είναι σε επίπεδο υπήρου και των τοπικών αγορών. Θα πιστεύω ότι θα δούμε ένα μείγμα λύσεων για αυτές τις αγορές όπου οι τοπικές λύσεις μπορούν να, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από άποψη κόστους και πάλι είναι μια προσωπική μου άποψη αυτή, όχι ως ε, Acer, ακόμα δεν έχω αναλάβει ε, στην Acer. Στο μέλλον λοιπόν θα δούμε λύσεις οι οποίες θα αφορούν το κόστος της υπηρεσίας που δεν θα είναι μόνο η παροχή ενέργειας αλλά και των ωφέλων ε, που ε, αφορούν και την παροχή ενέργειας. και τώρα όσον αφορά τον ε, ρόλο του σχεδιασμού και του συντονισμού. Ναι. Εκεί δεν είμαι τόσο σίγουρος, δεν έχω πολλή εμπειρία σχετικά με τις ε, προσπάθειες για την ε, αποθήκευση ε, και σύλληψη άνθρακα στην αρχή της διαδικασίας όμως τι είναι αυτό το οποίο θα προωθήσει την τεχνολογία θα είναι μια επαρκής τιμή για το διοξίδιο του άνθρακα. θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τιμή δεν είναι αρκετά υψηλή ακόμα. Όμως υπάρχουν πολλές προκλήσεις και όσον αφορά τις υποδομές. Και έτσι τίθεται το ερώτημα του ε, ποιος είναι ο ρόλος ε, ε, της ορθής ε, τιμολόγησης, όμως μπορεί να σταθεί από μόνη της όταν οι προκλήσεις είναι περισσότερες. Δεν νομίζω ότι ε, κάτι τέτοιο θα ισχύει. Βέβαια αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Τώρα όσον αφορά το PCI. Μελλοντικά μπορεί να εντοπίσουμε κόστος συγκεκριμένα για επενδύσεις όσον αφορά την ενέργεια και ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει ε, μια κυριαρχία ε, παρόχου. Υπάρχουν μόνο συγκεκριμένε περιοχές στην Ευρώπη ε, όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο, οπότε θα μειωθεί αυτό όσον αφορά τα προγράμματα για το φυσικό αέριο. Όμως όσον αφορά την εξάλληψη άνθρακα για το φυσικό αέριο, πιστεύω ότι εκεί ε, θα μπορεί να υπάρξουν ε, επενδύσεις ε, για τέτοιες υποδομές στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, εσείς μιλήσατε για τις τιμές ενέργειας που αποτελούν μια πρόκληση σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Η προσέγγιση που θα έχουμε ως υπηρεσία θα είναι ότι η πολιτική πολιτικές, ε, οι δημοσίες πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ε, φαινόμενο. Στο παρελθόν κάποιες από τις ε, παρεμβάσεις που γίνονται για να υποστηρίξουν αυτές τις θέσεις ήταν προσεγγίσεις για μια τιμή για όλους και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Πιο στοχευμένες παρεμβάσεις λοιπόν για την υποστήριξη της ε, τιμής, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό. Τώρα όσον αφορά ένα ερώτημα σχετικά με το πώς μπορούμε να περάσουμε από, το από τη θεωρία στην πράξη και το πώς βλέπω την υπηρεσία σε 10 χρόνια από τώρα και το πώς θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε το μήνυμα στους ε, πολίτες ε, θα έλεγα ότι αρχικά θα πρέπει οι ενεργειακέ αγορέ να λειτουργούν για τον καταναλωτή, ούτω ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, χαμηλότερο ε, κόστος και η ICE μπορεί να παίξει ένα ρόλο πάνω σε αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αγορέ θα είναι ανοιχτέ, ούτω ώστε νέοι καινοτόμοι παίκτε να μπορούν να παίξουν ένα ρόλο. Ε, δεν αφορά μονάχα ε, του όσου υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Και τρίτον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή ενσωμάτωση ως ε, έναν αποτελεσματικό τρόπο ε, για την εξάλληψη ε, εκπομπών άνθρακα στην οικονομία. Και αυτά λοιπόν είναι τα τρί, οι τρεις προτάσεις σχετικά με τους καταναλωτές και το πώς μπορείτε να το παρουσιάσετε στους καταναλωτές στις πατρίδες σας. Τώρα όσον αφορά ε, το Ταμείο της ε, Δίκαιης Μετάβασης, δύσκολη ερώτηση αυτή. Προσωπική μου θέση ότι ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης ε, το οποίο απλά θα ε, δίνει ε, επιδοτήσεις δεν πρόκειται να έχει, μία, δεν πρόκειται να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όμως ε, χρηματοδότηση που θα δίνεται για την βελτίωση και την αλλαγή των δεξιοτήτων τότε αυτό μπορεί να έχει αποτελέσματα όχι μονάχα όσον αφορά τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, αλλά και όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα το οποίο ε, εκτιμώ ιδιαιτέρως. Ε, στην δουλειά μου ταξιδεύω πολύ και πηγαίνω συχνά στην Ινδία, την Κίνα, Πηγαίνω για παράδειγμα λοιπόν σε ένα κινέζικο σούπερ μάρκετ ε, και εκεί βλέπω μια 80χρονη γυναίκα η οποία όχι μονάχα ψωνίζει και πληρώνει με το smartphone της ε, αλλά ε, συγκρίνει και τις τιμές διότι είναι 80 χρονών και τα κάνει όλα αυτά χωρίς να χρησιμοποιεί μετερετα Έχει τρομερές ψηφιακές δεξιότητες, είναι 80 χρονών. Το βρίσκω απίστευτο κάτι τέτοιο διότι ε, στην Ευρώπη κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο ούτε οι υποδομές για αυτό, αλλά ούτε και οι δεξιότητες και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Όσον αφορά το ε, τι μέλλον επιθυμούμε, αυτό δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά αφορά ε, και ε, το πώς πληρώνουμε, το πώς ψωνίζουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, αυτό θα βοηθήσει και στον τομέα της ενεργειακής ε, μετάβασης. Ε, αυτό ως μία πιο προσωπική απάντηση. Τώρα όσον αφορά τη σχέση με, την, τη σχέση με τα κράτη-μέλη και το ζήτημα του Nord Stream 2, η Acer λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθεί στενά ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί στις νομοθετικές αρχές ε, και τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα και όχι ακριβώς ε, να ε, μπει σε λεπτομέρειες που αφορούν πολιτικά ζητήματα. Αυτός πιστεύω ότι είναι ένας ε, καλός ε, τρόπος για να διατηρήσουμε την υποστήριξη που πρέπει να ε, δίνουμε και επίσης δεν είμαστε εξοπλισμένοι ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τέτοιων προγραμμάτων. Αυτό μπορούν καλύτερα να το κάνουν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί. κυρία Βάης, είχατε ένα ερώτημα σχετικά με τα μεγαλύτερα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε Πιστεύω ότι όπως είπε και ο κύριος Ποτότσνικ, η σύνδεση των αγορών και η καλύτερη χρήση των ε, διασύνδετών είναι ένα ε, θέμα και επίσης ε, το να δούμε που απαιτούνται ε, αγορές και να βοηθήσουμε εκεί πέρα και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε που ε, δεν είναι τόσο ε, σημαντικός ένας τέτοιος παράγοντας. Και ένα άλλο εμπόδιο, το οποίο δεν είναι τώρα εμπόδιο, αλλά μπορεί να γίνει μελλοντικά, να έχουμε μια πολύ ανοιχτή αγορά όπου έχουμε νέες εισόδους, με νέες προτάσεις, νέες καινοτομίες και να μην κλείσει αυτή η αγορά απλά και μόνο επειδή είναι μια ε, λύση. Αυτό θα είναι το σημαντικό. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή, όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να μην ε, γίνει πρόβλημα μελλοντικά. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι έχω απαντήσει ε, όλες τις ερωτήσεις και θα χαρώ να ακούσω τυχόν σχόλια. Εκτός μικροφώνου. Ε, δεν νομίζω ότι είναι η τελευταία μας ε, συνάντηση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή ε, αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Okay, then we move to the next point. Περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο Please, we have to start. Be seated. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Uh, Thank you, thank you very much. And, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο είναι η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού. 2018, για το 2018. Καλωσορίζω την κυρία Άννα Κολούτσι, διευθύντρια στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τα ζητήματα ενέργεια και περιβάλλοντο, ο κ. Γκυγιόμ Λογιό, ο οποίο είναι διευθυντή ε, για την ενημέρωση, την επικοινωνία και τα μίντια στην ίδια, Γενική ε, Διεύθυνση, και η κυρία Ντεκαστέλ, που είναι επικεφαλή ε, τη μονάδα. Σα καλώ να μα παρουσιάσετε αυτή την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού ιδιαίτερα βεβαίω ε, τις πτυχές που έχουν να κάνουν το ψηφιακό τομέα, τον τομέα της ενέργειας, να μας παρουσιάσετε το πού βρισκόμαστε, Κατευθείαν γραμμέ για την ενέργεια, για το περιβάλλον. Έχετε το λόγο, έχετε 10 λεπτά για αυτή την παρουσίαση, ο συνήθως μία ώρα συνολικά για τη συζήτηση. Παρακαλώ, δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει. Η κυρία Κολούτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την πολιτική ανταγωνισμού μας και την εφαρμογή στον τομέα της ενέργειας. Η ενέργεια βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας ε, γενικότερα από πλευρά ανταγωνισμού ο τομέας αυτός είναι, ε, εξαρτάται από την κρατική ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μεγάλη ρύθμιση του κλάδου, ε, μεγάλες εταιρείε είναι αυτέ που δεσπόζουν και τα κράτη-μέλη αποκλίνουν σημαντικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα του. Το περασμένο έτος, το 2018, το έτος δηλαδή αυτή τη έκθεση, αλλά και ε, κοντά στο τέλος της θητείας, η πολιτική ανταγωνισμού απάντησε θετικά ε, στις εκκλήσεις ή μια σωστή εφαρμογή του τομέα της ενέργειας που θα ε, συνεισφέρει στην Ενεργειακή Ένωση. Ο στόχος μας είναι να απαλείψουμε τα εμπόδια στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και να, να, πετύχουμε την αποθρακοποίηση εξασφαλίζοντας ε, την ε, ασφάλεια των εφοδιασμού και τη διασυνδεσιμότητα. Ε, ζητήματα αντιτράστ, κρατικών ενισχύσεων, στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα στα ζητήματα αντιτράστ, ε, αντιμετωπίζουμε μόνιμα προβλήματα με μεγάλη συγκέντρωση στις εθνικές αγορές. Περιορισμένη διασυνοριακή, περιορισμένος διασυνοριακός ανταγωνισμό και βεβαίως τα δίκτυα επίσης τα οποία ελέγχουν την αγορά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και που δείχνουν ε, τη δράση μας. Πρώτα είναι, πρώτα το θέμα της Gazprom που εγκρίθηκε το Μάιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια απόφαση που καθιστά ε, νομικώς δεσμευτική τη δέσμευση της Gazprom. Είναι βασικός προμηθευτής σε δεσπόρουσα θέση σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η Κομισιόν ανησυχούσε διότι η Gazprom ενδέχεται να είχε παραβιάσει τους κανόνες αντιτράστ ε, με μια στρατηγική κατακαιρματισμού των εθνικών αγορών και των αγορών φυσικού αερίου, δηλαδή σε 8 κράτη-μέλη. Και αυτό οδήγησε σε υψηλές τιμές φυσικού αερίου σε πέντε χώρες, τις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιβάλλοντας λοιπόν νομικά αυτές τις δεσμεύσεις στην Gazprom με μια σειρά από πολύ συγκεκριμένου κανόνε, αλλάξαμε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν η Gazprom και εξασφαλίσαμε ότι η αγορά φυσικού αερίου θα τυχαίνει των ίδιων ε, χαμηλών τιμών όπω στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η δεύτερη υπόθεση στην οποία θέλω να αναφερθώ έχει να κάνει με την ελεύθερη ροή ηλεκτρική συνέργεια μεταξύ Δανία και Γερμανία. Αυτή η απόφαση πάστηκε στα τέλη του προηγούμενου έτου και έχει να κάνει με την ΤΕΝΑΤ, τον, ε, το δίκτυο της Γερμανίας, τη σχετική επιχείρηση, και εκεί υπήρξε μια απόφαση δέσμευσης, δηλαδή δεσμευ... υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις ε, σε ό,τι αφορά αυτά που προσφέρει η ΤΕΝΑΤ. Εδώ είναι διαφορετικό το ζήτημα βέβαια. Ε, το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούσε ότι η ΤΕΝΕΤ συστηματικά περιόριζε τη δυνατότητα ε, της διασύνδεσης σε ηλεκτρικής ενέργειας που προχώταν από τις βόρειες χώρες δηλαδή από τη Δανία στην προκειμένη περίπτωση, που ήταν πιο φτηνές ε, προ τη Γερμανία. Παρεμπόδιζε δηλαδή την εξαγωγή αυτή τη ε, φτηνή ε, ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Γερμανία και αυτό βέβαια ε, οδηγούσε στο ότι οι Γερμανοί καταναλωτέ δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι πιο, πιο χαμηλές τιμές. αυτό που κάναμε ήταν και το blueprint στην πραγματικότητα της, ε, του κανονισμού για την ενέργεια ε, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των διασυνοριακών δυνατοτήτων ε, σε διασυνδέσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά για το αντιτράστ. Είχαμε και έντονη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Πέρυσι εγκρίναμε μια σειρά από προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και το συνδυασμό θέρμανσης ε, και ισχύω 21 προγράμματα εγκρίναμε και τα περισσότερα κράτη-μέλη πλέον έχουν λάβει σύμφωνη γνώμη σε ό,τι αφορά αυτά τα προγράμματα. Ταυτόχρονα χρειάστηκε να προσαρμόσουν του κανόνε του βέβαια και να ευθυγραμμιστούν αυτά τα προγράμματα με τι κρυπτέ γραμμέ και τι κρατικέ ενισχύσει ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό οδήγησε σε ένα χαμηλότερο κόστο για του καταναλωτέ. Έχουμε διαπιστώσει ότι στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, χάρη ε, στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων τη Ένωση, το κόστο των ανανεώσιμων πηγών, πηγών ενέργεια έχει μειωθεί κατά το ίμιση τα τελευταία χρόνια. Ένα άλλο τομέα δράση το 2018 έχει να κάνει με του μηχανισμό δυνατοτήτων. Όπω ξέρετε, ε, πρόκειται για τη δυνατότητα που δίνεται ε, να ανταμείβονται οι πάροχοι δυνατοτήτων ε, πέρα από τα έσοδα ε, από την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια ε, για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τις δυνατότητες ή να επενδύσουν και σε νέες δυνατότητες που είναι απαραίτητε ε, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεφοδιασμού. Εγκρίναμε 7 αποφάσεις, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία. Κάθε φορά η Κομισιόν αξιολόγησε το πρόγραμμα αυτά έτσι ώστε οι κανόνε κρατικών ενισχύσεων να γίνονται σεβαστοί αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ σημαντικό παράλληλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν ε, τα αριθμιστικά ζητήματα που υπήρχαν, τα αριθμιστικά κενά και να μην υπονομεύσει αυτό τα κίνητρα ε, για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να επενδύσουν σε νέες δυνατότητες. αυτό με φέρνει τώρα στις κατηδές γραμμές ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια. Όπως ε, είπατε και εσείς ε, νωρίτερα, θέλατε να σας πω κάτι σχετικά, διότι η δημόσια ενίσχυση στον τομέα αυτών διέπεται από τις κατηδές γραμμές που υπάρχουν από το 2014 και κατά την περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να επιτευχθεί η Ενεργειακή Ένωση μιας και εξασφαλίζουν ε, ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού χωρίς να περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα αυτό επιτρέπεται στον ορικό εμπόριο. Ε, ε, να σας εξηγήσω λίγο γιατί μεγέθη μιλάμε. όλα τα μέτρα, όλη η υποστήριξη που δίνουν τα κράτη-μέλη στην ενέργεια και στο περιβάλλον αποτελούν το, τη μισή στήριξη των συνολικών ενισχύσεων που δίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και σε αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε 241 αποφάσεις που αφορούν διάφορους τομείς, ε, ε, ενισχύσει ανανεώσιμες ποιες ενέργειες, ε, δημιουργία δυνατοτήτων, ε, ε μετριασμός των κοινωνικών ε, επιπτώσεων για το κλείσιμο μεταγωνιστικών επιχειρήσεων, κινητικότητα, ε, μεγάλο το εύρος όπως βλέπετε. Μόλις ξεκινήσαμε μια αξιολόγηση αυτών των κανόνων τον Ιανουάριο φέτος για να δούμε κατά πόσο οι κανόνες αυτοί είναι κατάλληλοι. Και αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε fitness check. Θα αναφερθεί σε λίγο τώρα η συνάδελφος σε αυτό. Για μας είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε και για το Green Deal που ανακοίνωσε η νέα πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, να προσαρμόσουμε τι νέε κρατικέ γραμμέ ε, στο πρόσφατο πακέτο για την καθαρή ενέργεια που εγκρίθηκε πέρυσι, να προσαρμόσουμε τι κρατικέ γραμμέ και στη τεχνολογική πρόοδο και τι δυνατότητε που υπάρχουν. Ε, η Don Deal για την αποθήκευση, για το υδρογόνο, πολύ σημαντικά στοιχεία για την απανθρακοποίηση ε, και να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και τις εξελίξεις στην αγορά στον τομέα της ενέργειας. Παραδείγματο χάρη είναι το γεγονός ότι έχουμε ε, χαμηλή ε, κινητικότητα εκπομπών. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας καθώς θα προχωρούμε στην αξιολόγηση αυτή, στο fitness check. Θα δώσω τώρα το λόγο στην συνά, στον συνάδελφο, στον κύριο Βαντεκαστέλ, που θα αναφερθεί ακριβώς στο fitness check. Well, we have revised the... Έχουμε αναθεωρήσει τους περισσότερες ε, κρατικές νομοθεσίες από το 2004 μέχρι το 2014 στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού δηλαδή των κρατικών σχετικών διατάξεων και εξάλλου αυτές οι νομοθεσίες εκπίπτουν εκπνέουν οι περισσότερες του χρόνου. Επίσης έχουμε κάνει και ε, έλεγχο αντιστοίχησης για την τομήνυμης, για τις περιφερειακές κατευθύνες γραμμές για ενισχύσεις το πλαίσιο σημαντικών project κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, τις κατευθύνσεις γραμμές για τη χρηματοδότηση κινδύνου, τις κατευθύνσεις γραμμές για την αεροπλοεία, για την ενέργεια, ε, για τις, ε, τον κατασκευαστικό τομέα και επίσης έχουμε και ένα, ε, έχουμε κατευθύνσεις γραμμές και για τους σιδηροδρόμους αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πολύ μεγάλο πακέτο δηλαδή. Έχουμε γενικά προβεί σε διαβούλευση που ολοκληρώθηκε φέτος τον Ιούλιο. Έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα σύνολα κανόνων ρυθμίσεων που ολοκληρώθηκαν επίσης ε, τον Ιούλιο. Για το IPCI και τα project καινού ευρωπαϊκού συμφέροντος έχουμε στείλει ερωτηματολόγιο το οποίο παρατάθηκε μέχρι πρόσφατα, το τέλος του Οκτωβρίου, 21 Οκτωβρίου και παράλληλα έχουμε μια, μια σειρά μελετών που γίνονται για αυτούς τους διαφορούς τομείς ε, σε σχέση με το κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις στην αεροπλοεία έχουμε προχωρήσει πολύ και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του έτους. Έχουμε δύο άλλες μελέτες που αφορούν ε, την ενέργεια ε, και το περιβάλλον και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη που μάλλον θα συνεχιστούν μέχρι τον επόμενο χρόνο. Για να σας δώσω μια προκαταρκτική ενημέρωση για αυτό το έλεγχο <coughs> κατάστασης που κοιτά προς το παρελθόν για το κατά πόσο δηλαδή οι κανόνες έχουν λειτουργήσει σωστά και αν, θα, και αν χρησιμεύουν, εξακολουθούν να χρησιμεύουν. Η πρώτη αντίδραση είναι πως αυτοί οι κανόνες εν γέννη φαίνεται να λειτουργούν ε, καλά. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά από τεχνικές παρατηρήσεις που έχουν ε, γίνει και που πρέπει να εξεταστούν πιο στενά ε, όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα αναθεωρήσουμε ή όχι κάποιους από αυτούς τους κανόνες. Πρακτικά λοιπόν τα επόμενα βήματα είναι ότι εργαζόμαστε για τη συνόψιση και τη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων από όλες αυτές τις μελέτες. Αυτά θα καταγραφούν σε ένα έγγραφο που ε, εκθέτει την κατάσταση προόδου και θα περάσει και από το Συμβούλιο ε, Εποπτείας. Ε, και μετά θα δούμε και θα λάβουμε ε, απόφαση γιατί αν χρειάζονται κάποιες τεχνικές προσαρμογές ή αν χρειάζεται πλήρης ε, μεταρρύθμιση και αναθεώρηση κάποιων κανονισμών. Εάν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται τέτοια εκβάθρον αλλαγή, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες επιλογές τις οποίες θα πρέπει και να δοκιμάσουμε. Και μετά θα ακολουθήσει αυτή καθ' αυτή η νομοθετική διαδικασία. Αυτή είναι μια γενική εικόνα λοιπόν για το που βρισκόμαστε με αυτό το έλεγχο καταλληλότητας. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Λοριό να ενημερώσει για το υπόλοιπο κομμάτι. Ε, καλησπέρα σας, ονομάζομαι Κυριό Λοριό. Είμαι υπεύθυνο της διεύθυνση για την επιχειρησιακή επιβολή των κανόνων ε, ανταγωνισμού και αντιδράστη, δηλαδή κατάχρηση κυρίαρχης θέσης, έλεγχος συγχωνεύσεων στην ε, αγορά της, κοινο... της τεχνολογίας της πληροφορίας που καλύπτει μεγάλες εταιρείες αλλά και μικρές εταιρείες και θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γενική εικόνα για τις δραστηριότητες επιβολής που έχουμε κάνει το τελευταίο χρόνο. Επίσης, ποιες είναι οι συζητήσεις, πολιτικές συζητήσεις που ξεκίνησαν με βάση τις εκθέσεις των ειδικών συμβούλων που είχε καλέσει η Επίτροπος Φεσχάγκερ να ε, ε, ασχοληθούν με την ψηφιακή σφαίρα. Βέβαια, οι ψηφιακές αγορές είναι ευρύτερε από τη δική μου ε, δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, γιατί πλέον η ψηφιακή τεχνολογία μπαίνει παντού. Τώρα, για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού σε αυτό το ψηφιακέ αγορέ ε, ICT, τις επιγραμμικές αγορέ, υπήρξαν κάποιες εργασίες γνωστέ που καλύπτουν διάφορες υποθέσεις που είχαμε και κυρίως ενάντια στην Google, κατά της Google. Είχαμε και άλλε περιοχές επιβολή ειδικά το τομέα της ε, επιγραμμικής διανομής. πολύ ε, ε, ιδιαίτερο θέμα είναι ο ανταγωνισμός ε, των ψηφιακών πλατφορμών, όχι μόνο την Google αλλά και άλλες πλατφόρμες. Μια τρίτη απόφαση λήφθη το 2019 κατά της Google για μια διαφορετική αγορά που είναι ειδική αγορά επιγραμμικής διαφήμισης και έρευνας αλλά και διαμεσολάβησης όπου η Κομισιόν εξέτασε την Google για ορισμένες πρακτικές αποκλειστικότητας για τις διαφημιστικές αγορές δηλαδή πρακτικές διαφορετικού τύπου από αυτές που είχαμε ε, εντοπίσει ας πούμε για την Google Android που υιοθετήθηκε το 2018 και σχετιζόταν με διαφορετική αγορά αλλά κατά βάση πρόκειται για κινητή τηλεφωνία και τη σχετική πλατφόρμα με διάφορα θέματα που αφορούσαν ε, το χρόνο, τον ε, κερματισμό και την αποκλειστικότητα και έπειτα την απόφαση Google Shopping που υιοθετήθηκε το 2017 και φορούσε πάλι μια ακόμα άλλη πρακτική. Έχουμε δει δηλαδή μια μεγάλη ποικιλία από καταχρήσεις, τις οποίες έχουμε εντοπίσει, έχουμε υιοθετήσει διάφορες αποφάσεις, οι οποίες όπως ίσως γνωρίζετε τώρα είναι στο δικαστήριο. Υπάρχει μεγάλη προετοιμασία, προετοιμάζουν τις ακροάσεις, τις ακροαματικές διαδικασίες, είναι πολύ μεγάλες υποθέσεις με πολλά τμήματα, με πολλά μέρη ε, που κυρίως υποστηρίζουν την Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Άλλες ερευνές, ορισμένες εξ αυτών έχουν δημοσιευθεί, όπως ας πούμε η έρευνα που ξεκινήσαμε πέρσι το καλοκαίρι κατά της Amazon, Όσον αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με αγορές, πρόκειται για δημόσιες πληροφορίες, δημοσιευμένες, αλλά η έρευνα συνεχίζεται ώστε να κατανοήσουμε κατά πόσο η Amazon έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί δεδομένα τρίτων μερών που πολλούν στην ίδια αυτή την πλατφόρμα με στόχο να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην ε, αγορά λιανικών πωλήσεων, όπου η Amazon έχει ε, ε, πωλήσεις. Επίσης, άλλη απόφαση αφορούσε τα ηλεκτρονικά βιβλία. Και άλλη υπόθεση αφορά την Apple και το Spotify και γίνονται και άλλες έρευνες που δεν μπορώ ακόμα να σχολιάσω. Ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Όλες αυτές οι υποθέσεις λοιπόν αφορούν διαφορετικού είδους πρακτικές και διαφορετικές αγορές. Έχουμε να κάνουμε με ζητήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει αρκετά νωρίς, ας πούμε... Σε κάποιες αγορές υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο ρόλο που παίζει μια πλατφόρμα και την τοποθέτησή της σε μια συγκεκριμένη αγορά και τη δραστηριότητά της σε μια άλλη αγορά. Και εκεί τίθενται πολύ περίπλοκα ζητήματα, τα οποία καταρχάς πρέπει να εντοπίσουμε, να περιγράψουμε και μετά να δούμε κατά πόσο επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό είναι θέμα βέβαια το οποίο απασχολεί όλες τις εθνικές ε, ε, αρχές ανταγωνισμού και την Κομισιόν. Και ήταν άλλωστε αυτός και ο στόχος της έκθεσης ε, ε, ε, των ειδικών συμβούλων, η οποία εξέθεσε κάποιους προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστούμε την επιβολή antitrust. Πώς δηλαδή από την μια πλευρά θα διατηρηθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις πλατφόρμες, σε περίπτωση δηλαδή που οι αγορές, γιατί θέλουμε οι αγορές να παραμείνουν χώροι ανοιχτοί σε διάφορες πλατφόρμες, αλλά και περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισμός γίνεται μέσα στην ίδια την πλατφόρμα, όπου η ίδια πλατφόρμα δηλαδή μπορεί κατά κάποιο τρόπο να λειτουργήσει ως ρυθμιστής εντό εισαγωγικών και να εξασφαλίσει ότι είναι ισότιμο το πεδίο για όλους, εφόσον μία πλατφόρμα μπορεί να είναι ο χώρος ε, στον οποίο ανταγωνίζονται διάφοροι ψηφιακοί ε, φορείς. Όλα αυτά ήταν χρήσιμα λοιπόν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι ε, πρακτικές γίνονται ε, σε ένα σύστημα όπου υπάρχει δυνατότητα <laughs> για τα δεδομένα, ας πούμε, βλέπουμε διάφορες αγορές όπου η αξία των δεδομένων έχει πολύ σημαντικό ρόλο, είτε στο να έχουν πλονέκτημα, ανταγωνιστικό, είτε οι ανταγωνιστές να μην μπορούν να ανταγωνιστούν επίση ώρε και αυτό έχει εξεταστεί στο πλαίσιο μεγάλων υποθέσεων, όπως ας πούμε ε, στην υπόθεση Microsoft, όπου η Κομισιόν ζήτησε διαλειτουργικότητα για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός πάνω στην ίδια πλατφόρμα. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζονται όχι μόνο για να ενημερωθούν οι αρμόδιε αρχέ, αλλά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό η Κομισιόν να μπορεί να κερδίσει αυτέ τι υποθέσει του επόμενου μήνε και χρόνια, ώστε να μπορέσει να ε, προστατεύει τον ανταγωνισμό και να συνεχίζει την ε, στεναρή επιβολή όλων των νομοθετημάτων. Πέρα από τις πλατφόρμες είδαμε και τον τομέα της επιγραμμικής διανομής που επίσης ακολουθεί την τομεακή έρευνα που κάναμε με το e-commerce όπου μπορούμε να δούμε ότι επίσης υπάρχουν κάποιες πρακτικές περιορισμένες ανάμεσα στους προμηθευτές και στους διανομής, ειδικά όταν πρόκειται για τον περιορισμό των πωλήσεων εντός της ενιαίας αγοράς, δηλαδή συνοριακού τύπου ε, περιορισμοί. Η Κομισιόν έχει συνεχίσει φέτος να επιβάλλει τα άρθρα 1 και 1.02 όταν βλέπει ότι υπάρχουν ε, ρυθμίσεις που εμποδίζουν από τον καταναλωτή, τον καταναλωτή από το να εκμεταλλευτεί την ενιαία αγορά και να μπορέσει να αγοράσει επιγραμμικά από διαφορετικούς προμηθευτές εντός της Ένωσης και να ωφεληθεί από την ενιαία αγορά. Υπήρξαν τέτοιες υποθέσεις, ας πούμε, όσον αφορά την αδειοδότηση εμπορικών προϊόντων, όπου οι αγορές δεν ήταν πολύ μεγάλες ως αξία, αλλά ως προηγούμενο είχαν μεγάλη αξία. Ήταν πολύ σημαντικές αποφάσεις που δείχνουν ότι η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει ότι ο ανταγωνισμός θα καλύπτει και τις, τους διασυνοριακούς περιορισμούς. Και όταν ξέρεις ότι η Κομισιόν θα αναθεωρήσει τις, ε, τις ε, κατευθύνες γραμμές για την κατακόρυφη ε, διανομή το 2020, τότε σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι, οι θύνοντες για τη λήψη αποφάσεων είναι πολύ σημαντικές αυτές οι κατευθύνες γραμμές για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις αγορές. Τέλος, να πω δύο λόγια για το είδος της επιβολής που γίνεται στις ε, αγορές ε, υψηλής τεχνολογίας, γιατί είχαμε υποθέσεις στις αγορές διαφόρων ε, τσίπ. όπου είδαμε συγκεκριμένη εταιρεία να έχει καταχραστεί την κυρίαρχή της θέσης, ασκώντας μία ε, αρπακτική πολιτική όσον αφορά τα τσιπ. Ε, αυτή η υπόθεση έχει λήξει τον περασμένο Ιούλιο. Επίσης, η Κομισιόν 18 χρόνια μετά από την υιοθέτηση απόφαση, τέτοιες απόφασης που ελήφθη δηλαδή το 2001, η Κομισιόν έλαβε ένα ενδιάμεσο μέτρο ενάντια στην πρώτη κόμμα, δηλαδή υπόθεση κατάχρησης κυρίαρχης θέσης, όπου αποφάσισε να ε, διατάξει την Broadcom να σταματήσει πρακτικές αποκλειστικότητας και μόχλευσης σε κάποιες αγοράς, αγορές ε, chip, ε, όπου μπορεί να συγκεκριμένοι κατασκευαστές, μόντεμ ή τέτοιου είδους ε, ε, προϊόντων αναγκάζονται να, να κλείσουν λόγω αυτών των πρακτικών. Και αυτή ήταν πολύ σημαντική απόφαση, γιατί δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τι δυνατότητε που έχουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να επιβάλλουμε ε, την προστασία του ανταγωνισμού, όταν βλέπουμε δηλαδή ότι μπορεί έτσι να προκληθεί ένα επανόρθωτη βλάβη. Πολύ σημαντικό λοιπόν για την Επίτροπο να δείξει ότι όταν και μπορούμε και έχουμε τα στοιχεία είμαστε ε, αποφασισμένοι να υιοθετήσουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Νομίζω πως έτσι έχετε μια γενική εικόνα, αλλά αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. And, uh, so after this presentation we... Μετά από αυτή την ε, παρουσίαση μπορούμε να περάσουμε στην συζήτηση από το ΕΛΚ η κυρία Βάις. Ο, κύριο ο κύριος ε, Ζήλινσεν στο τελευταίο του ε, σχόλιο προηγουμένως είπε ότι στο μέλλον θα πρέπει να ε, προσέξουμε ο ανταγωνισμός ε, στην αγορά ενέργειας θα πρέπει να είναι ε, ανοιχτός ε, και ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Πώς λοιπόν μπορεί η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό να συνεισφέρει στη, στο, στη φιλόδοξη πράσινη συμφωνία και πώς τα εργαλεία για τον ανταγωνισμό θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στην πράσινη μετάβαση για την Ευρώπη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσουμε ε, να ανασχεδιάσουμε ε, τον ε, τομέα ανταγωνισμού. Δεν έχουμε κάποιον από τους σοσιαλδημοκράτες, από το Ρινιού; Ευχαριστώ πολύ. αναφέρεται ότι η Επιτροπή συνεχίζει και ε, προωθεί μία ε, ανταγωνιστική αγορά και ε, προς όφελος των καταναλωτών. Επίσης προσπαθεί να δημιουργήσει δίκαιες πρακτικές το θέμα της ε, διαφάνειας ε, θα πρέπει να αποτελέσει βάση για τα κράτη-μέλη. Όμως, σε ορισμένες χώρες ο ανταγωνισμός ε, αντιμετωπίζει στρεβλώσεις, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους καταναλωτές. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έριξε τις τιμές αερίου ε, κάτι το οποίο σήμαινε φθηνότερε τιμές για τους καταναλωτέ, αλλά κινδύνευσε να οδηγήσει σε χρεοκοπία τη επιχειρήση. με τις ε, τιμές να πέφτουν από το 2014 αυτή τη στιγμή ένας ε, ε καταναλωτή στην Ουγγαρία πληρώνει περισσότερο από ό,τι θα πλήρωνε άμα ήταν ελεύθερη η αγορά να ρυθμίσει τις τιμές. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί ε, ακριβές ε, διαδικασίες κατά το οποίο παραπλανεί τους καταναλωτές και σε αυτό το πλαίσιο συμφωνείται ότι οι αρχές της Ενεργειακής Ένωσης αλλά και της διαφάνειας και του δίκαιου ανταγωνισμού δεν συμφωνούν με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην Ουγγαρία. Τώρα για τους πράσινους. θα επικεντρωθώ στο ζήτημα της ενεργειακής μεταφοράς, ε, μετάβασης ε, σε μια, σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς τις ε, εκπομπές Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας. Δεν είναι μονάχα να επιλύσουμε τις ε, ε, ρυθμιστικές, ε, τα ρυθμιστικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να βοηθήσουμε τις κοινότητες και να ανοίξουμε την ενεργειακή αγορά για τους μικρότερους ε, για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή με την αξιολόγηση της ε, λέει ότι θα πρέπει να εκπληρωθούν τα, προετοι... τα ώστε να προωθηθεί περαιτέρω ε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας επίσης τις εκπομπές και αθώς επίσης και τις συνέπειες που θα έχει στο περιβάλλον. Αυτά είναι θύματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως είναι για παράδειγμα την ε, μείωση του τεχνολογικού κόστος, ε, την, ε, το φθηνό κεφάλαιο, καθώς επίσης και σταθερές τιμές όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, ε, θα πρέπει να μειώσουμε, να μειώσουμε τις τιμές στην αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές, να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική ε, εφαρμογή των ε, εργαλείων που θα προωθούν την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές Πολλά προαπαιτούμενα λοιπόν, αυτά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα ήθελα από πλευρά σας να μας πείτε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς επίσης και για την αγορά που θα ε, εκπληρώνουν τους ε, στόχους ε, για το 2050 και επίσης θα βοηθήσουν προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος από το IND. Από το ECR. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τομιτσόφσκι. Θα ήθελα να να ακούσα σχόλια σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον ενεργειακό τομέα Δεν είναι ε, δυνατό λοιπόν να, εξυγχρονι... να εξυγχρονίσουμε όλες τις εγκαταστάσεις ε, θέρμανσης, ε, για παράδειγμα, που εκεί παρατηρούνται μεγάλες απώλειες ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές λοιπόν Ε, μπορεί να σημαίνουν ε, ε, εξοικονόμηση ενέργειας και γι' αυτό τον λόγο σκέφτεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανονισμούς σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις πάνω σε αυτό το θέμα τους ώστε να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα των υδροελεκτρικών ε, επιχειρήσεων. Έχει στείλει μια επιστολή η Κομισιόν σε σε 8 κράτη-μέλη, Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Γαλλία, δύο μια πρωτοπερική επιστολή όπου λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν σέβονται την οδηγία του 2014 για τι διορτικέ ε, άδειε. Εμεί η Γαλλία μάλλον θίγεται ιδιαίτερα εδώ, διότι ε, παρα, υπήρξε παράταση κάποιων αδειών χωρίς διαγωνισμούς. Ε, υπάρχουν διαγωνισμοί για 150 άδειες που λήγουν το 2023. Είναι όμως παράλογο το να ανοίξουμε στον ανταγωνισμό την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι παράλογο για την ασφάλεια των χρηστών, για την ασφάλεια του εφοδιασμού, μιας και ο κάθε αδειούχος θα ακολουθεί ε, τους οικονομικούς τους στόχους και όχι τους στόχους αξιοπιστίας και ασφάλεια του συστήματος. Βάζουμε σε ανταγωνισμό ε, ορισμένες φορές ε, ε, με παράλογο τρόπο εταιρείε που είναι στην ίδια, ε, στην ίδια περιοχή. Ε, οικολογικά είναι προβληματικό το, το, ζήτημα. Οικονομικά επίσης, μια και θα αυξηθεί η τιμή για τον καταναλωτή. Οπότε οι ερωτήσεις μου είναι απλές. Είμαστε στην εποχή του Green Deal και της δίκαιης μετάβασης. Η οδηγία του 2014 θα τροποποιηθεί έτσι ώστε ο τομέας της ηλεκτρικής να μην, να μην υπόκειται στον ανταγωνισμό. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τουλάχιστον τους ιστορικούς ε, παρόχους ως ε, παρόχους μιας υπηρεσίας καθολικής ε, ε, χρησιμότητας ε, και να μην υπάρχει έτσι ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να θέσω ερώτημα. Γιατί εν μέρει είναι και προσωπικό το ερώτημα. Αναφερθήκατε ε, στην ε, Gazprom και την ε, θέση της στην ενεργειακή αγορά. Το ερώτημα μου δεν είναι ιδιαίτερα τεχνικό. Για ποιο λόγο η Επιτροπή είναι τόσο αβοήθητη όσον αφορά την Gazprom. Αν αναλογιστούμε την απόφαση του 2016 για τον ε, Σολίνα Όπεν ε, απερίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους γνωστούς λόγους ε, και τώρα έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε προβλήματα με την εφαρμογή σχετικά με τα όσα αποφασίσαμε και κατά την προηγούμενη θετία του Κοινοβουλίου όσον αφορά την Gazprom. Έχω τις προσωπικές μου αφιβολίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό θα είναι κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Για ποιο λόγο λοιπόν αντιμετωπίζουμε αυτή την εταιρεία η οποία είναι ένα ε, πρόβλημα και στους τομείς τους, του ανταγωνισμού. Για ποιο λόγο λοιπόν ε, ε, την αντιμετωπίζουμε τόσο ήπια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ μπορείτε να απαντήσετε. Θα ξεκινήσω με την ε, πρώτη ερώτηση της κυρίας Βάης. σχετικά με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες ε, για τον ανταγωνισμό θα βοηθήσουν στην παράδοση της Πράσινης Συμφωνίας και ότι ε, ο ανοιχτός και ευέλικτος ανταγωνισμός θα μπορέσει να βοηθήσει στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης. Όπως είπα, υπάρχουν ε, δύο ε, δράσεις, δύο πλευρές δράσης. Από τη μία έχουμε την εφαρμογή και από την άλλη την δράση πολιτικής όσον αφορά την επιβολή. Η Επιτροπή έχει επιδιώξει τα τελευταία χρόνια ε, μια ε, πολύ αυστηρή πολιτική ε, εφαρμογή για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η αγορά θα λειτουργεί σωστά, διότι αυτή θα είναι η πρώτη βάση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα παραδοθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο απόψης κόστους για τον καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά τώρα θα πρέπει να δούμε τα εργαλεία πολιτικής τα οποία έχουμε στον ε, τομέα της ε, πολιτικής ε, ανταγωνισμού. Όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον, έχουμε τους, την νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στο παρελθόν. Για παράδειγμα, μπορέσαμε να μειώσουμε το κόστος των ανανεώσιμων ε, και επίσης ε, στο fitness ε, check που διεξάγαμε το, οι πρώτες πληροφορίες που λάβαμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ότι αναγνωρίζουν πως τα εργαλεία αυτά πραγματικά έχουν λειτουργήσει και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το θετικό στοιχείο θα διατηρηθεί. Ταυτόχρονα όμως θα, θα πρέπει να εξετάσουμε το τι θα σημαίνει η Πράσινη Συμφωνία για την οικονομία και για τους καταναλωτές και εκεί θα πρέπει ε, αυτό να φαίνεται στους, ε, στην νομοθεσία και οι κανόνες ε, δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα για τις νέες τεχνολογίες όπως είναι για παράδειγμα το υδρογόνο, η καθαρή κινητικότητα, η αποθήκευση. Λάβαμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις φόρτισης, όμως αυτό, αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συνθήκης και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το προσαρμόσουμε σε νέα ένα νέο νομοθετικό εργαλείο, ούτως ώστε να μας βοηθήσει στη διαδικασία εξάλληψης εκπομπών και τους στόχους που έχουμε θέσει για μέχρι το 2050. Τώρα, επειδή το ερώτημα αυτό συνδεόταν ε, και ε, με αυτό εδώ το ερώτημα του κυρίου Νίστο από τους ε, πράσινους, ε, αναρωτηθήκατε σχετικά με το πώς ε, ε, η, κρατική νομοθεσία θα ε, συνάδει με τους στόχους μας, ενώ ταυτόχρονα θα είμαστε αποτελεσματικοί από άποψη κόστους είναι ένας από τους στόχους τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν κάνουμε τις αξιολογήσεις και τις αναθεωρήσεις των κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις η αποτελεσματικότητα κόστους ε, θα διασφαλίζει ότι οι επιδοτήσεις που θα δίνουν τα ε, κράτη-μέλη θα είναι αναλογικές ε, και αυτή είναι μία από τις ανησυχίες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι Άλλα στοιχεία όπως είναι η ανταγωνιστικότητα επίσης θα λαμβάνονται υπόψη. Ναι, μερικές φορές μπορεί να υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο στοιχείων. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Τώρα αναφέρθηκε το θέμα του κόστους ε, και, το, ε, και η περίπτωση της Ουγγαρίας. Για να μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την ε, ενέργεια θα πρέπει όλοι οι παράγοντες της αγοράς να ακολουθούν τις ε, τους κανόνες, ε, ε, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός ε, για τους, διότι αν έχουμε περισσότερο από έναν πάροχο θα ανταγωνίζονται για την παροχή αλλά και για τις τιμές και αυτό είναι το οποίο προσπαθεί να επιτυχεί η πολιτική μας. Αυτό αναφέρεται και στην οδηγία για τον ηλεκτρισμό που υιοθετήθηκε στο πακέτο καθαρής, στη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Ε, σε κάποιες χώρες μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις τώρα όσον αφορά την ελεύθερη τιμολόγηση. Έτσι λοιπόν για ευάλωτους ε, καταναλωτές ε, θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε μια ρύθμιση ε, της τιμής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε εξέχουσες περιπτώσεις αυτό εφόσον δεν επηρεάζει την αγορά χονδρικής θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την ρύθμιση της τιμολόγησης όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται το ότι δεν θα έχουμε πολλαπλές επιδοτήσεις ή ότι θα έχουμε τιμές κάτω από το κόστος. Έτσι λοιπόν από τη μία πλευρά έχουμε μια νομοθετική προστασία η οποία προσφέρει στα κράτη-μέλη την ε, ε, κατευθυντήριο σχετικά με το πώς ε, θα μπορεί να γίνεται η ρύθμιση της τιμολόγησης και από την άλλη πλευρά έχουμε την πολιτική εφαρμογής μέσω του ανταγωνισμού όπου και εκεί εξετάζουμε το αν η ρύθμιση της μολόγησης ιδιαίτερως σε επίπεδο χονδρικής θα μπορούσε να ε, προσφέρει πλεονεκτήματα σε ορισμένες ε, ε, βιομηχανίες εις βάρος άλλων και εν τέλει και εις βάρος του καταναλωτή. Τώρα η Επιτροπή έχει αποστείλει επιστολή σε διάφορα ε, κράτη-μέλη ε, όσον αφορά ε, τα, εργα... τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, μεταξύ αυτών και η Γαλλία. Όταν εξετάζουμε την κατάσταση στην Γαλλία, εφόσον αυτό ήταν το ερώτημα που ητέθη, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι παραχωρήσεις έχουν ε, αφορούν ε, μονάχα μία εντότητα χωρίς ε, ανταγωνισμό και θα έλεγα ότι λειτουργούν με τις ίδιες περιουσίες για τους καταναλωτές με τις καλύτερες δυνατές τιμές για αυτούς και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί όταν έχουμε τις ε, παραχωρήσεις και τις συμφωνίες στον τομέα του ανταγωνισμού. Ότι, τα, ότι αυτό το οποίο ότι ο καλύτερος ε, πάροχος ε, μπορεί να είναι υπεύθυνος για αυτές τις παραχωρήσεις ή οι επιχειρήσει οι οποίε ε, μπορούν να χειριστούν αυτέ τι παραχωρήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο από άποψη κόστου ε, θα μπορούν επίση να εξυπηρετούν του ε, καταναλωτέ και τα κράτη-μέλη μπορούν να το κάνουν αυτό προ όφελο του καταναλωτή. Οι ίδιοι πάροχοι λοιπόν που είναι υπεύθυνοι για αυτό αυτές τις υπηρεσίες στη Γαλλία ενδιαφέρονται και ε, για την ε, δραστηριοποίησή τους ε, και σε άλλες αγορές και πιστεύουμε ότι αυτό για τη Γαλλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλά ωφέλη εν τέλει για τους καταναλωτές. Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα σας κύριε Πρόεδρε όσον αφορά την Gazprom και την απόφαση για την Gazprom για ποιο λόγο είμαστε τόσο βοήθητοι απέναντι στην Gazprom Ναι, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την απόφαση που λάβαμε πέρσι, η οποία ήταν μια δέσμευση, αυτό το οποίο βλέπουμε όταν λαμβάνουμε ε, αποφάσεις τέτοιες μας επιτρέπουν να διασφαλίσουμε ότι συγκεκριμένες δράσεις θα ληφθούν από ε, την ε, συγκεκριμένη ανάληψη υποχρέωσης και οι δεσμεύσεις ε, που έγιναν ε, νομικά δεσμευτικές ε, θα αλλάξουν την συμπεριφορά της Gazprom σε αυτά τα κράτη-μέλη. Οι δεσμεύσεις αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα να γίνει μια σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν σε, άλλες, σε άλλα κράτη-μέλη και αυτό ε, λοιπόν αποτελεί μια πολύ ισχυρή δέσμευση και η ε, Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή τους από την ε, Gazprom. Θα έλεγα λοιπόν ότι από τη δικιά μας εμπειρία οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές και ένα σημαντικό διορθωτικό μέτρο στην αγορά και η παρέμβαση της Επιτροπής ε, δεν σταματά στην υιοθέτηση, αλλά στη συνέχεια ακολουθεί και η παρακολούθηση, ούτως ώστε οι δεσμεύσεις αυτές όντως να εφαρμόζονται. Ελπίζω λοιπόν ε, να έχω καλύψει όλες τις ερωτήσεις, παρόλα αυτά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις εάν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Εάν όχι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για την παρουσίαση, τις απαντήσεις. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο της διάταξης. Ε, τώρα περνάμε στα διάφορα πρέπει να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στις 4 Δεκεμβρίου. Εδώ στις Βρυξέλλες. Κοινή συνεδρίαση με μια άλλη επιτροπή. Επίσης, η συνεδρία των συντονιστών θα ξεκινήσει στις 5 και μισή. Είμαι λίγο κουρασμένο, συγγνώμη. Yeah.